Καλησπέρα σα λέει ο Πρόεδρος. Καλώς ορίσατε συνάδελφοι και καθίστε. Να αρχίσουμε. δεν έχουν έρθει και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Βέβαια είναι Δευτέρα, τσαγκαρό Δευτέρα, αλλά ας αρχίσουμε. Γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Το πρώτο εκ των οποίων είναι η έγκριση της σημερινής σα διάταξης, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις. Το σχέδιο αυτής, όπως σας έχει διανεμηθεί, εγκρίνεται. Η διερμηνία γίνεται από όλες τις, ε, προς όλες τις από όλες τις γλώσσες, εκτός από κελτικά, λετωνικά, λιθωνικά και φιλανδικά και τώρα τις ε, ανακοινώσεις του Προέδρου όσον αφορά τις εφαρμοστικές και κατεξοδότηση πράξεις. Κατόπιν τη εγγράφου διαδικασία τη Δευτέρα 12 του 19, οι συντονιστέ συμφώνησαν με πλειοψηφία να ζητήσουν από τον Πρόεδρο να απευθύνει επιστολή σε Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να του ε, ενημερώνει για την καινούργια προθεσμία της ε, διαδικασίας ελέγχου σε σχέση με τον κανονισμό αυτών του Συμβουλίου για το εσωτερικό Ταμείο Ασφαλείας και είχαμε πει ότι έχουμε δύο εφαρμοστικές πράξεις ε, που αποφασίστηκε στις 26 Νοεμβρίου που αφορούν την Europol και την Interpol της βάσης δεδομένων όπως επίσης και την διαλειτουργικότητα για σύνορα και βίζες. Η προθεσμία για υποβολή ενστάσεων ορίστηκε η δεκάτη δωδεκάτου. Αύριο το μεσημέρι συγκεκριμένα. Αυτό όσον αφορά τις και τώρα προχωρούμε στα θέματα ουσίας για σήμερα. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, EDPB. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι προβλέπεται η, η παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων από τον Αντρία Γέλεν που είναι ο πρόεδρος του EDPB. Η οποία, κυρία Γέλνικ, θα μας πει για αυτή τη νέα υπηρεσία η οποία αντικαθιστά την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 που υπήρχε παραδοσιακά. Τώρα υπάρχει αυτό το συμβούλιο, αυτή η υπηρεσία. Σας ευχαριστούμε κυρία Γέλνεκ που ήρθατε. Που ήρθατε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Θα ακούσουμε την παρουσίασή σας και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει περιθώριο για συζήτηση αμέσως μετά. Δώσουμε το λόγο σε όποιον συνάδελφο θέλει να υποβάλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Έχετε 10 λεπτά. Άντε 12. Εάν θέλετε. Και μετά όμως έχουμε κάποια άλλα ζητήματα, κάποια ζητήματα νομοθετικά. Αλλά και συζήτηση με τον νέο Επίτροπο για Ιστορικές Υποθέσεις, την κυρία Γιωχάνσον η οποία θα είναι μαζί μα στι 4 παρατέταρτο. Οπότε ελπίζουμε να τηρήσουμε τα χρονικά πλαίσια. Για αυτό το πρώτο μα θέμα που είναι από τι 3 μέχρι τι 4 ε, παρατέταρτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και ευχαριστώ όλα τα μέλη τη Επιτροπή σα για την πρόσκληση και έχω την τιμή να σας παρουσιάσω ε, αυτό το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να σας πω τι είναι το EDPB. Είναι μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή υπηρεσία που βοηθά στο να υπάρχει ε, συνεπής συμμόρφωση της προστασίας των δεδομένων σε όλη την Ένωση και έτσι να έχουμε τη συνεργασία ε, των αρμοδίων αρχών. Έχουμε σε δύο υπηρεσίες για αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ του Συμβουλίου Προστασίας και της ε, εποπτικής αρχής. Οπότε θα πρέπει να συγχαρώ τον ε, νέο επόπτη, τον κύριο Γεβαρόφσκι, που πρέπει να βλέπει πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων από τα θεσμικά όργανα, το πώς όλοι γνωρίζετε. Και το Συμβουλίο μας θεσπίστηκε από τον ε, Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων για να μπορούμε να έχουμε μια συνεπή εφαρμογή του σχετικού κανονισμού από τι εθνικέ εποπτικέ ε, αρχές για επιχειρήσεις όποιον άλλο διέπεται από τη χρήση των δεδομένων, αλλά και τι μας αρχές. Έχουμε επομένω τις εθνικές ε, αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι χώρε ΕΖΕΣ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία και EDPS. Οπότε η τοποθέτησή μας έχει σχέση και με το ότι έχουμε και την γραμματεία του Συμβουλίου που υπάγεται κατευθείαν στον στην Πρόεδρο. Επίσης είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο των αποφάσεων εθνικών οργάνων. Ούτε είναι ρυθμιστικό όργανο ή αρχείο δεν αντικαθιστά τις αντίστοιχες εθνικές αρχές. Οι υποπτικές αρχές είναι εθνικές, ανεξάρτητες, κοντά στον πολίτη και έχουν αρμοδιότητες και μέσα να εφαρμόσουν τον νόμο και μπορούν να επιβάλλουν και χρηματικές ποινές. Η υπηρεσία μας επομένω δεν είναι δευτεροβάθμιο όργανο των εθνικών αποφάσεων, οι οποίες ε, μπορούν να κρυφθούν από τις εθνικές δικαστικές αρχές. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και ελέγχει τις ε, εθνικές διατάξεις σε σχέση με τον γενικό κανονισμό. Εμείς βοηθούμε. Τώρα, η αποστολή μας. Έχουμε τρεις βασικές αρμοδιότητες. Γενικά θέτουμε κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το δίκαιο προστασίας δεδομένων της κοινότητας προς τις εθνικές αρχές, να υπάρχει ερμηνεία συνέπειας. Επίσης ε, προσπαθούμε να υπάρχει συνέπεια όσον αφορά τις ε, αποφάσεις των εθνικών αρχών. Και έτσι οι εθνικέ νομοθεσίε να εφαρμόζονται με μειώνφο τρόπο και επίση έχουμε και συμβουλευτικό ρόλο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποια θέματα που έχουν σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προτινόμενη νέα νομοθεσία στην Ένωση. Ιδίω όταν αυτή έχει ιδιαίτερα σημασία για την προστασία των σχετικών δεδομένων και για κάποια απόφαση που σχετίζεται με τρίτη χώρα. Σας είπα ότι έχουμε ως αρμοδιότητα τις καθημερινές γραμμές. Μέχρι τώρα έχουμε 16 τέτοιες και άλλες 8 από τότε που άρχισε να ισχύει ο Γενικός Κανονισμός των στις 25 Μαΐου του 18. Μετά την έγκριση αυτού του σχεδίου κατευθυντηρίων υπευλήθησαν σε διαβούλευση πριν ολοκληρωθούν. Πέντε κατευθυντήρες έχουν ολοκληρωθεί μέσω των διαβουλεύσεων και άλλες τρεις τώρα βρίσκονται στη διαδικασία της διαβούλευσης. Και τώρα είναι ένα από τα πιο επίμαχα ζητήματα του γενικού κανονισμού τις αποφάσεις και την συνέπεια για να εξασφαλιστεί η συνέπεια για την εφαρμογή του κανονισμού η υπηρεσία μας μπορεί να λάβει δεσμευτικές αποφάσεις οι οποίες απευθύνονται σε εθνικές υποφτικές αρχές. Είμαστε ο φορέας επίλυσης διαφορών όταν υπάρχουν τέτοιες διαφορές μεταξύ εθνικών αρχών που συνεργάζονται για κάποια υπόθεση διασυνοριακή. Μέχρι τώρα δεν έτυχε κάτι τέτοιο σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού. Εκδίδουμε γνωμοδοτήσεις για κάποια θέματα που θεωρούνται ότι έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Οι πολιτικές αρχές δεν μπορούν να αποφασίσουν πριν διαβουλευθούν με την υπηρεσία μας. Μέχρι ότου εμείς γνωμοδοτήσουμε προς αυτές. Αυτό ισχύ με κάποιους κώδικες διοντολογίας, πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις προστασίας δεδομένων. Έχουμε γνωμοδοτήσει σχετικό 41 φορές μέχρι τώρα. Όπως προανέφερα, γνωμοδοτούμε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποτύπων συμβουλής, να σου πω κάποια ε, παραδείγματα, φερειπίν για την ε, απόφαση καταλληλότητας, ε, όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ Ιαπωνίας, τον κανονισμό για το e-privacy, προστασία ηλεκτρονική ιδιωτικού βίου, ε, την ασπίδα προστασία ιδιωτικού βίου, επίσης το FATCA, ε, το φορολογικό της Ηνωμένης Πολιτείας και άλλα. Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού. Αυτό το έχουν οι εθνικές εποπτικές αρχές. Για να δούμε τώρα περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Οι εποπτικές αρχές έχουν περισσότερες αρμοδιότητες με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού. Και τώρα μπορούν να επιβάλλουν χρηματικές ποινές μέχρι 10 έως 20 εκατομμύρια ευρώ σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ανάλογα με την παράβαση. Επίσης μπορούν να επιπλήξουν ή να προειδοποιήσουν. Και πρέπει η θέση του Πρόεδρου του οργανισμού μας να αντιστοιχεί σε Εθνική Εποπτική Αρχή. Προβλέπεται επίση σύστημα συνεργασίας αυτών των εθνικών ευρωπαϊκών αρχών και υπάρχει ένα κεντρικό σημείο επαφής. Και αυτό το λέμε μηχανισμός μόνο απευθυντική θηρίδα. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Βλέπετε τώρα ένα σχήμα για το πώς λειτουργεί αυτός ο οργανισμός. Βλέπουμε ότι την κυρίως αρμόδια αρχή Επίση, υπάρχουν εθνικοί κανόνες και έτσι μοιράζονται πληροφορίε με άλλες ε, εθνικές αρχές. Η ε, κυρίως ε, αρμοδιά υπηρεσία είναι εκεί που υπάρχει η έδρα κάποια εταιρεία. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε κοινοποιείται ένα σχέδιο απόφασης στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και αν δεν υπάρχουν ενστάσει για το σχέδιο κειμένου, τότε η αρμόδια αποπτική αρχή συμφωνεί με το σχεδίο απόφασης. Αυτή είναι η φάση της συνεργασίας. Και βλέπετε εδώ ότι ο μηχανισμός ε, συνέπειας λειτουργεί όταν υπάρχει κάποια ένσταση, κάποια διαφωνία. Οπότε και τότε εμείς λειτουργούμε ως υπηρεσία επίλυσης διαφοράς. Και οι υποπτικές αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη την απόφασή μας ή στην τελική απόφαση που αφορά τα ε, μέρη τα οποία έχουν την αντιδικία. Άρα είπαμε ότι αυτό ισχύει μόνο όταν υπάρχει κάποια διαφωνία. Τώρα αυτός ο μηχανισμός εθνικής θηρίδας είναι κάποια βελτίωση για τις επιχειρήσεις σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς ιδέα εταιρείε έχουν μόνο μία εποπτική αρχή με την οποία να συνομιλήσουν και όχι πολύ περισσότερες. Αυτό είναι πιο απλό και πιο φτηνό για τι επιχειρήσει τη Ένωση. Οι δε εποπτικέ αρχέ, εξασφαλίζουν την συνέπεια στι αποφάσει και στο τέλο τη διαδικασία και τη διαδρομή υπάρχει μία απόφαση που ισχύει διασυνοριακά άσχετα από το πόσε είναι οι συναρμόδιε εποπτικέ αρχέ. Τώρα, για ε, να έχετε μια άποψη για το πώς, τι ισχύει, έχουμε 766 τέτοιες περιπτώσεις συνεργασίας που έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό μήτρο. Αυτό από 4 Δεκεμβρίου 470 είναι υποθέσεις μόνο ευθυνικής θηρίδας και από αυτές τις υποθέσεις ήδη οι 74 ήδη διέπονται από κάποια τελική απόφαση. Για αυτές τις διασυνοριακές υποθέσεις η πλατφόρμα του IMI δεν φτιάχνει ότι το δική μας υπηρεσία ούτε για, τις προστασίες, για την προστασία δεδομένων, αλλά προσαρμόστηκε είναι το σύστημα πληροφοριών ιστορικής αγοράς για να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών των αρμοδιών αρχών και έτσι μπορούν οι υπηρεσίε να μπουν σε ένα σύστημα, αλλά και αυτό το σύστημα προσαρμόστηκε για τι δικέ μα ανάγκε. Οπότε η υπηρεσία μα ε, δεν παρεμβαίνει ε, όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας σε κρατημέλη ή για την διεκπαιρέωση των καταγγελιών και φτάνει σε εμά το θέμα όταν υπάρχει κάποια διαφορά, κάποια προστιβή όπως σας προείπα. Και έχουμε πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία στο σύστημα IMI. Όπως γνωρίζετε, γιατί το έχουμε δημοσίευσει αυτό στις αρχές του έτους, έχουμε ένα αυστηρό και σφιχτό πρόγραμμα για το 2019-2020. Οι εποπτικές αρχές έχουν υψηλό φόρτο εργασίας και εθνικό και διασυνοριακό, αλλά και σε επίπεδο ε, η TPP της ε, δικής μας, EDPP μάλλον. Ε, πάνω από 12 είναι κατευθυντήριες γραμμές για να καταλαβαίνουν καλύτερα και να ε, εφαρμόζουν καλύτερα το γενικό κανονισμό και με μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή. Η πρώτη τέτοια άσκηση για την προστασία δεδομένων ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία. Και τώρα προχωρούμε για να εγκρίνουμε γνωμοδοτήσεις για το BCR και στάνταρ ε, ε, ρήτρε της συμβάσει, ε, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επαφίενται σε δοκιμασμένα ένομα μέσα. Και έχουμε πάρα πολλή δουλειά με τους μηχανισμούς ε, πιστοποίησης και κώδικες ε, δεοντολογίες που είναι και άλλα εργαλεία αυτά λόγω δοσίας. Θα εξακολουθήσουμε να παίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο συμβουλεύοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σημαντικά ζητήματα προστασίας δεδομένων. Και εκτός από την καθημερινή δουλειά θέλουμε να συνεισφέρουμε και στη διεθνή συζήτηση που γίνεται για την προστασία δεδομένων και να συνεργαστούμε με τέτοιες αρχές παγκοσμίω. Τώρα κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση αυτό το θέμα, καθώς επίσης και είναι προτεραιότητα ε, των πολιτικών. Η προστασία των δεδομένων πραγματικά ε, συζητείται παντού στον κόσμο, έχει γίνει viral. Ε, θα βλέπετε εδώ στο χάρτη πόσο αυξάνεται η σημασία της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι πάνω από 100 πλέον οι χώρες παγκοσμίως που έχουν σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ η υπηρεσία μας είναι υπέρ της περαιτέρω σύγκληση αυτής της νομοθεσίας παγκοσμίω. Στόχο έχουμε να φτάσουμε σε ένα βαθμό συμβατότητας ή σύγκληση μεταξύ ε, των διεθνών συστημάτων προστασίας δεδομένων για να έχουν αυξημένα επίπεδα ε, εμπιστοσύνη ή ε, επιχειρήσεις και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως χώρας. Ο νέος γενικός κανονισμός με τους σύγχρονους κανόνες εξασφαλίζει ισχυρή προστασία ε, των προσωπικών δεδομένων. Εμείς θέλουμε η Ευρώπη να έχει παρουσία και επιρροή ε, στη διεθνή συζήτηση που γίνεται για την προαγωγή υψηλού επίπεδου προστασίας. Για να γίνει όμως αυτό και να αντιμετωπίσουμε το φόρτο εργασίας που έχουμε και τις προκλήσεις, χρειαζόμαστε Μάλιστα, ξέρετε ότι συνεδριάζουμε 11 φορές ε, το χρόνο ε, στις Βρυξέλλες και εν ώψη αυτών των συνεδριάσεων έχουμε πάρα πολλές συνεδριάσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Πάνω από 100 τέτοιες συνεδριάσεις είχαμε το τελευταίο 18 μήνο. Ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθούμε σε αυτό το έργο μας είναι ε, να έχουμε σωστή στελέχωση. Ιδιαίτερα αν έχετε υπόψη ότι ε, ο Ευρωπαίος νομοθέτης μας ανέθεσε και το συντονισμό των ε, συστημάτων πληροφορικής. Είναι και Eurojust, το σύστημα VIS, ε, το σύστημα SIS, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενημέρωση για τα ποινικά μητρώα και ενημέρωση για τις άδειε ε, ταξιδίων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ε, επιπλέον φόρτο και εμεί και οι γραμματείε μα. πέρα από τη δουλειά που έχουμε ήδη να κάνουμε. Επίσης θα παρακολουθήσουμε στενά ε, οποιοδήποτε νέο ρόλο μα ανατεθεί στα πλαίσια ενό κανονισμού πούμε, για την ιδιωτικότητα στον χώρο. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σα Έχουμε πολλού ρόλου και αναλυτικό και επιμελητίας και ε, είναι και κόμβο επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων εποπτικών αρχών αλλά και με εξωτερικούς ενδιαφερομένους. Πρόσφατα μάθαμε ότι ο προπολογισμό για το 2020 εγκρίθηκε και θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τα μέλη της Επιτροπής σας για την υποστήριξή σας στις ε, διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω λέγοντας ότι στην υπηρεσία μας συνεργαζόμαστε με τον επόπτη προστασίας και με τις εθνικές εποπτικές αρχές πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε κοινό στόχο να ε, εφαρμόζονται τα θεμελιά δικαιώματα ε, των Ευρωπαίων πολιτών ε, με πάντα μεγάλη ισορροπία των εθνικών με τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Είναι περίπλοκο αυτό το εγχείρημα και χρειάζεται ε, τους απαραίτητους πόρους για να πετύχει. Εμείς είμαστε ρυθμιστική αρχή και θεωρούμε ότι οι συνομοθέτες είναι βασικοί συνομιλητές και εταίροι μας, γιατί το θέμα μας το έχουν ψηλά στην πολιτική τους ατζέντα ως προτεραιότητα, για να προστατεύονται αποτελεσματικά ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ιδίως το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ Γέλνεκ. Data Protection Board, EDPB αγαπητέ Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Και ευχαριστούμε και την Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων που έκανε αυτή τη παρουσίαση για τη σημαντική αυτή καινοτομία με τη θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι ένα σημαντικό νομοθέτημα στα πλαίσια της δέσμης ε, της νομοθετικής, στην οποία ε, ήμασταν προσιλωμένοι στην προπερασμένη θητεία, από το 2009 μέχρι το 2014 και καταφέραμε στην επόμενη ε, θητεία, το 2014 και έλεγα στην κυρία Γέλινεκ ότι το όνομά της πραγματικά μας θυμίζει πολλά εμάς που είμαστε παλιοί και έχουμε σπουδάσει και νομική. Ε, και έχουμε αυτή τη νομική σκέψη. Γιατί ήταν ο καθηγητής Γκέρκ Γέλινεκ και ο γιος του, Βάλτερ Γέλινεκ, που κυριάρχησαν στη διαμόρφωση ε, ε, του Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου και είχαν τεράστια επιρροή στο γερμανικό και αυστριακό δημόσιο ο δόκτωρ Γέλινεκ ήταν καθοριστικός καθώς συνέταξε το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης που γιορτάζει τώρα την εκατοστή επέτειο από το 1999-2019. Ε, ε, και σε μικρότερο βαθμό επηρέασε πολύ και την τσεχική και την ε,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 Πρώτον, από πλευρά σας υπάρχει κάτι που έχετε την αίσθηση ότι στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρειάζεται κάποια βελτίωση ή κάτι άλλο να προσθέσουμε. Δεύτερη ερώτηση. Μιλήσατε για τις ε, ε, στάνταρ ρήτρες ε, στις συμβάσεις, αλλά κάτι που δεν άκουσα να είπατε. Έχετε κανένα πρότυπο για ένα τέτοιο κώδικα δεοντολογίας έχετε αναπτύξει κανένα κείμενο ε, έτσι πρότυπο ε, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη ε, και οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να συμφωνήσουν. Και τρίτον, η υπηρεσία σας εστιάζει μόνο στην προστασία των πολιτικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή μήπως αναπτύσσετε και κάποια πράγματα εν ώψη της καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης ε, να ε, οδηγούν σε κάποιες λύσεις. Δηλαδή, ασχολείστε μόνο με την προστασία των δεδομένων ή εξετάζετε και θέσεις και δυνατότητες για το πώς μπορεί κανείς να φτάσει σε κάποιους στόχους χωρίς να παραβιάζει τελικά τα προσωπικά δεδομένα. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Σίπελ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κυρία Γέλινεκ. Δύο τομεί θέλω να αναφέρω. Όπως είπατε και εσείς, οι πόροι και ε, οι εθνικοί, εθνικές αρμόδιες αρχές και οι ευρωπαϊκές είπατε ότι δεν είναι επαρκής και με βάση τον γενικό κανονισμό η προσοχή, το ενδιαφέρον και εμείς ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία των δεδομένων για την προστασία της ιδιωτικότητας, της δημοκρατίας, των θεωρητών δικαιωμάτων. είναι ένα αυτόνομο αριθμό ερωτήσεων, καταγγελίων κτλ. Σε εσά το Συμβούλιο ε, Προσωπικών ε, ε, Δεδομένων υπάρχει επαρκή στελέχωση, υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες και Και το δεύτερο, αυτή η μοναπαθητική θηρίδα που αναφέρατε και είπατε ότι συνιστά σημαντική βελτίωση, θα συμφωνήσω καταρχήν μαζί σας προς αυτό. Ακούγονται όμως ε, φήμες ε, ότι σε ό,τι αφορά ε, το Ιρλανδικό γραφείο υπάρχουν πολλές καταγγελίες, έχουν να κάνουν το Facebook και τα και στην πράξη τελικά πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι καταγγελίες, γιατί είναι επιβαρημένες οι Ιρλανδικές αρχές. Πρόκειται άλλωστε για πολύπλοκες καταγγελίες και αναφορές. Υπάρχει συνεργασία, ότι δηλαδή να τα αρμοδιότητες σε κάποια στάδια της διαδικασία σε άλλους φορείς, σε άλλες αρχές. Ή πιστεύετε ότι χρειάζονται βελτιώσεις ή αλλαγές στον κοινωνισμό προς αυτό. Τώρα για το Ρινιούλιο Πρόεδρος. Ποιος θα έχει το λόγο, η κυρία Ιντεβέλτ ή ο κύριος Μπράι. Γιατί είπατε κυρία Ζίπελ, κατάλαβες κύριε Πρόεδρε, με τα χαράς. Ε, πάντα ε, ε, είμαστε ανοιχτοί σε νέα mail. Ναι, θα μιλήσω εγώ στον Ίστρια. Κυρία Γέλνικ, σας ευχαριστούμε. Έχω καμιά δύο ερωτήσεις που έρχονται να προσθεθούν σε ερωτήσεις των συναδέλφων, που είναι και αυτές πάρα πολύ σωστές και εύστοχε. Ήδη απευθύνθηκα σε εσά εγγράφο για τα θέματα τη διαφάνεια προκαιρού και ιδίω για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών. Μέχρι στιγμή δεν πήρα κάποια πλήρη απάντηση, αν μπορώ να το πω έτσι, και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον προτίθεστε να δημοσιεύετε τα πρακτικά και σε ποια εξαίρεση αναφερθήκατε στον κανονισμό περί διαφάνειας για να δικαιολογήσετε τη μη διαμοσιοποίηση, Γιατί ειλικρινά νομίζω ότι με τη δημοσιοποίηση η οργάνωσή σας θα καταστεί πιο ισχυρή, δεν θα αποδυναμωθεί. Δεύτερον, για την επιβολή. Ε, τεταμένως μας εξηγήσατε πώς λειτουργεί. Αν κάνουμε όμω ένα βήμα πίσω και το δούμε το θέμα με τα μάτια των πολιτών, ναι, μεν έχουμε την καλύτερη νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας στον κόσμο, δεν είναι όμως ε, επαρκής πρακτική εφαρμογή. Σε εκατομμύρια δολάρια πρόστιμα ε, επιβάλλονται στη ΣΥΠΑ, στην Ευρώπη αυτό δεν το βλέπουμε. Γιατί είμαστε τόσο αδύναμοι πάνω από ένα και μισό, ενάμιση χρόνο έχει τεθεί σε ισχύ ο γενικός κανονισμός. Δεν θα έπρεπε να έχουμε αναλάβει δράση. Και ένα άλλο ερώτημα που σας είχα επίση απευθύνει γράφωση ήταν το PNR, η συμφωνία μας με τον Καναδά. Το δικαστήριο το ευρωπαϊκό λέει ότι ο Καναδάς ή οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να ε, βάσει τα δεδομένα ε, PNR μόνο σε χώρες ε, που ε, προσφέρουν επαρκή προστασία και στην ερώτησή μου λέτε ότι προσυπογράφεται ε, τις απόψεις της Ομάδας Εργασίας 29, το άρθρο 29, ότι αυτό αφορά είπα. δηλαδή οποιαδήποτε διαβίωση δεδομένων μεταξύ Καναδά ας πούμε και ΕΠΑ ή οποιασδήποτε άλλη χώρας και ΕΠΑ θεωρείται παράνομη. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι θα κάνετε με αυτό. Δεν αρκεί να έχει κανείς μια άποψη για κάτι, αλλά πρέπει και να παρεμβαίνει, να αναλαμβάνει δράση. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν, ευχαριστώ. Πρόεδρο, εμεί ευχαριστούμε για του πράσινου. Ο κύριο Μπράιερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τρει ερωτήσει έχω. Η πρώτη αφορά την επιβολή. Υπάρχουν κάποιες κοινέ δράσεις τις οποίες ε, προτείνετε ή έχετε ήδη δρομολογήσει καλό θα ήταν ε, η επιβολή να γίνεται συντονισμένα μεταξύ κρατών μελών. Και το δεύτερο ερώτημα, οι Ιρλανδικές αρχές, ο ε, Ιρλανδικός επόπτης, ε, η επεξεργασία, η διαδικτυακή είναι ένα θέμα στο οποίο εστιάζουν και οι πόροι δεν επαρκούν και από ό,τι άκουσα έχουν ζητήσει ε, υποστήριξη και σε συγκεκριμένους τομείς από άλλες αρχές. Οι Ιρλανδοί, πώς ε, προτείνετε να λύσετε το πρόβλημα λιματικής εφαρμογής ε, για την Ιρλανδία. Και τρίτον, υποχρεωτική διακράτηση δεδομένων Ξεκάθαρα έχει πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι δεν μπορούν να κρατηθούν, να φυλαχθούν όλες οι ανακοινώσεις, τα στοιχεία ε, δεδομένων που αφορούν την, ε, τον εντοπισμό όλων των πολιτών. Όμως, πολλά κράτη εισάγουν νέα ε, νομοσχέδια σχετικά. Το Συμβούλιο δεν πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη στάση προς αυτό για να μην συμβαίνει δηλαδή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. ID. Υπάρχει κάποιο πρόθυμος ή από το CCR, κάποιος που να θέλει να μιλήσει. Αν όχι, κυρία Ντέιλεκ, μέρο τη Ευχαριστώ, Πρόεδρε για την Ιρλανδική Αρχή, για τον ελληνικό Επόπτη, Επόπτη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιε αποφάσεις που αναμένονται από την Ιρλανδική Υπηρεσία μετά τι έρευνε που έκαναν το καλοκαίρι για Facebook ιδίω και για WhatsApp. Και έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία Ουσιαστικά είναι οι πρώτες αποφάσεις μετά την θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού ε, και έχουμε και τις ε, άλλες αποφάσεις ό,τι αφορά τις ε, τεχνολογικές εταιρείε από τις ΕΠΑ. Νομίζω ότι οι υπόπτες κάνουν καλή δουλειά, δεν νομίζω ότι κολλησιεργούν, αλλά είναι και σε δύσκολη θέση γιατί πολλά διακυβεύονται εδώ. Γνωρίζουμε ότι για, τη, το Facebook και τις άλλες υποθέσεις οι δικηγόροι έχουν ε, κάνει πολλές ερωτήσεις για την ε, ανταλλαγή δυνητικά ευαίσθητων πληροφοριών μας από τις άλλες χώρες, άρα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα δούμε. Το ερώτημά μου είναι, ε, όπως και άλλοι συνάδελφοι έθεσαν, το τι μπορεί να κάνει το Συμβούλιο για να στηρίξει τον επόπτη, τον Ελλανδό, σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία. Αυτό είναι το βασικό μέλημα και η βασική μου ανησυχία αυτή τη στιγμή. Πρώτα, ευχαριστώ. κάποιο άλλος. Θέλει κάτι να πει για αυτό το νέο οργανισμό. Board replacing the former... Κυρία Πιούρικ, έχετε το λόγο σας. Mr. Chair, um... As demonstrated... Σπούρικ, Μια έρευνα που έγινε στην Πολωνία φέτος έδειξε ότι το 54% των απαντώντων έχουν ε, αμφιβολίες για το Τα πόσον ε, υπάρχει έρευνα συμμόρφωσης ικανοποιητική. Σε μεγάλες οργανώσεις μπορεί τα ποσοστά είναι καλύτερα, αλλά το 59% των μεγάλων εταιριών αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ερμηνεία του καγενικού κανονισμού. Φαντάστε τι, Φανταστείτε τι προβλήματα θα αντιμετωπίζουν πιο μικρές επιχειρήσεις. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν το Συμβούλιο σας ερεύνησε ή θα ερευνήσει τι εκπαιδευτικέ δραστηριότητε τη Κομισιόν, τις επικοινωνικές δραστηριότητες Κομισιόν Κρατών Μελών, αν έγιναν και αν έγιναν, τι ήταν αυτέ για την σωστή εφαρμογή του γενικού κανονισμού, γιατί υπάρχει ελπίση συμμετοχή, ε, εφαρμογή και αυτό επηρεάζει, όπω ήθιστε, του ηλικιωμένου, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και τους λιγότερο ε, εύπορους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, τώρα υπάρχει κανένα άλλο ή όχι. Κυρία Κινίτσι, Φάτσα Λοπούρε. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε και την κυρία Γέλινεκ που ήρθε εδώ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας και για την εισήγησή σας και για τη δουλειά της υπηρεσίας σας. Για ό,τι κάνατε και θα συνεχίσετε να κάνετε. Μία ερώτηση τώρα συγκεκριμένη σε σχέση με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι. Συνέχεια μας είπε η κυρία Σπούρεκ για κάποια θέματα, ε, για κάποιους τέλος πάντων που είναι πιο ευάλωτοι και ενώ τους ε, ανηλίκους, γιατί υπάρχουν κάποια ανήλικοι στις πιο τρυφερές ηλικίε που έρχονται σε επαφή με καινούργια τεχνολογία και την πληροφορική. Και σας ερωτώ, στο γενικό κανονισμό τονίζεται με συγκεκριμένο τρόπο η προστασία που πρέπει να απολάβουν για τα προσωπικά δεδομένα οι ανήλικοι. Γιατί δεν έχουν τόσο συνέστηση των κινδύνων και βέβαια ούτε τα δικαιώματά τους δεν ξέρουν. Για πέστε μας. Ο φορέας σας τι μέτρα προτίθεται να λάβει ούτως ώστε να υλοποιήσει αυτή την προβλεπόμενη προστασία των ανηλίκων και συγκεκριμένα Πώς έχετε περιβάλλει προστασία τους ε, ανήλικους σε σχέση με την κώδικα διοντολογίας ε, που θέλετε να θεσπιστεί μαζί με άλλα θεσμικά όργανα. Τι γίνεται επίσης με τα άλλα δικαιώματα που βλέπει ο κανονισμός. Ε, κατά πόσον κάποιος μπορεί να σβήσει τα του που τα έχει εισαγάγει στο δίκτυο τι γίνεται με τους ε, νέους και με τους ακόμη πιο νέους. Πώς είναι δυνατόν αυτό το δικαίωμα να το απολάβουν. Θα πρέπει στα διάφορα website να προβλέπετε ε, με σαφήνεια και συντομία οι δε αρχές να πρέπει να μπορούν να υποπτεύσουν αυτή, την, αυτή τη ρύθμιση και έτσι να καταπολεμηθεί το bullying. Ο πρόεδρος και τώρα η σκητάλη στο Προεδρείο, η δε κυρία θα απαντήσει τις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί. Όσο πιο σύντομα τα πείτε, τόσο καλύτερα γιατί προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος για κάθε σημείο και έπεται το επόμενο, η επόμενη προσκεκλημένη αλλά και η Επίτροπος κατά τις 4.30. Ήδη, ήδη έχουμε καθυστερήσει από ό,τι βλέπω, λέει η κυρία Γίλνες, να σας τα πω συντόμως, ή στα γερμανικά προς τους Γερμανούς που ερώτησαν. Κύριε Φως, κύριε Βουλευτά, μιλήσατε για ε, κάποια επαναξεργασία που θα χρειαστεί ο Γενικός Κανονισμός ε, θα γίνει μια αξιολόγηση, θα συμμετέχουν πολύ ενδιαφερόμενοι, πρώτα τα κράτη, δεύτερον οι αρμόδιες αρχές, οι κρατικές εποπτικές αρχές και η δική μας υπηρεσία. Ο γενικός κανονισμός είναι ένας συμβιβασμός που προέκυψε μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και ένας πολύ καλός συμβιβασμός. Φυσικά πάντα χωράει βελτίωση, αλλά δεν είναι υποχρεωτική αυτή. Ε, για το κείμενο του κανονισμού. Αυτό που χωράει βελτίωση και θα μπορούσαμε ε, να το κάνουμε, αλλά αποφάσισαν διαφορετικά τα κράτη-μέλη, ε, είναι να υπάρχουν διοικητικοί κανόνες για την εφαρμογή κοινή. Αυτό θα διευκόλυνε πολύ τα πράγματα, αλλά δεν έχει να κάνει με το γενικό κανονισμό και ισχύει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις για τις τυποποιημένες ρήτρε ε, κάποιες συμβάσεις ε, Υπάρχουν κάποιε τέτοιε στάνταρ που έχει βγάλει ο Δανό υπόπτη και μπορούν και οι άλλοι να προσανατολιστούν σε αυτό. Ε, Επίση, ρωτήσατε αν εργαζόμαστε Προ την κατεύθυνση να επιτυχάνουμε κάποιους στόχους χωρίς να παραβιάζουμε τον κανονισμό, τον γενικό κανονισμό. Υπάρχει δυνατότητα αυτό, ε, αλλά για τους εθνικούς επόπτες, τις εθνικές εποπτικές αυτές. Όταν μια εταιρεία καλείται να κάνει μελέτη αντικτύπου ως προς τα προσωπικά δεδομένα και δεν λαμβάνει υπόψη όλους τους κινδύνους, μπορεί να επέμβει ο επόπτης ε, και να έχει συμβουλευτικό ρόλο ε, σε εθνικό επίπεδο. Και συμβαίνει επίσης. Αυτό είναι πολύ καλό αυτό το μέσο του συγκεκριμένου Γενικού Κανονισμού Προστασίας για την κυρία Σίπελ. Μιλήσατε για τους πόρους των Εθνικών Εποπτικών Αρχών ε, και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της δικής μας υπηρεσίας. Σας ευχαρίστησα ήδη την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την υποστήριξη για τους δικούς μας πόρους, ε, τον προπολογισμό και έχει, υπάρχει δυνατότητα του χρόνου να προσλάβουμε πέντε νομικούς στη γραμματεία μας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δεν είναι τόσο ρόδινο όμως τα πράγματα παντού στις εθνικές εποπτικές αρχές. Τα τέσσερα πέμπτα θα έλεγα των αρχών αυτών είτε είναι υποστελεχωμένα είτε είναι υποχρηματοδοτούμενα. Αλλά αυτό είναι ζήτημα των εθνικών Προπολογισμών και στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαπιστώνει εάν επαρκούν οι πόροι ή όχι. Μπορεί να είστε βέβαιοι ότι πάντα διαπραγματεύονται οι επόπτες προστασίας ε, με τις κυβερνήσεις του και στην Αυστρία συμβαίνει αυτό. Έχουν αυξηθεί τα αιτήματα, έχετε δίκιο. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Σε εμάς δεκαπλασιάστηκε ο φόρτος εργασίας και οι καταγγελίες στην Αυστρία και όχι μόνο. Φυσικά ε, το προσωπικό δεν το έχουμε ή μόνο απευθυντική ε, θηρίδα για την Ιρλανδία. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και κάποιες διαδρομές. Είναι περίπλοκες οι διαδικασίες αυτοί και όχι μόνο στην Ιρλανδία και παντού μέχρι να βρουν το δρόμο μέχρι τον επόπτη. Απλώς έχουν άλλη απήχηση και στην κοινή γνώμη αλλά και γενικότερα. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι πλήττονται, που πλήττονται κιόλας. Ε, η συνεργασία ε, είναι πολύ αγαστή, αλλά είπα και προηγουμένως για ε, τις εθνικές διαδικασίες πολλές εποπτικές αρχές έχουν δεμένα τα χέρια τους. Στην Τσεχία, την Αυστρία και την Ιταλία υπάρχουν προθεσμίες για λήψη αποφάσεων και στην Ισπανία νομίζω. Στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν προθεσμίες, ούτε στη Γερμανία. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλιώς δεν θα υπήρχε ε, η δυνατότητα να αποφασίσει κανεί εν ευθέτω χρόνο. Τώρα η συνεργασία, όχι μόνο με την Ιρλανδική Εποπτική Αρχή, αλλά και με τις υπόλοιπες, είναι πολύ καλή. Φυσικά και η ανταλλαγή των πληροφοριών και της ενημέρωσης ποικίλει χρονικά από χώρα σε χώρα. Διαπίστωση είναι αυτό, δεν είναι αξιολογική κρίση. Πάντως όλοι ε, φροντίζουν πολύ προσεκτικά, ε, γιατί όλοι θα πρέπει να ε, επαγρυπνούμε αυστηρά και να περιμένουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται αποφάσει κατά τον οποίο σίγουρα ορισμένοι θα προσφύγουν θα πρέπει να ε, στέκουν και στα δικαστήρια. Στα αγγλικά τώρα ε, για την κυρία Νιτφέλτ, σε ό,τι αφορά τα πρακτικά μας και τη διαφάνεια. Τα είπαμε. Νομίζω στην τελευταία σύνοδο. Τώρα αξιολογούμε με ποιο τρόπο θα τα πάμε καλύτερα. Είπαμε ότι θέλουμε διαφάνεια και σωστή βιώνει τον εξώ κόσμο αλλά να μην θίγεται η λήψη αποφάσεων και να μην θίγονται οι διαφαθμισμένες διαδικασίες, όπως επίσης έρευνες και διερευνήσεις. Μα γίνεται ανταλλαγή πολλών πληροφοριών και θα πρέπει να προσέξουμε τι θα δημοσιοποιείτε. Να είστε σίγουροι ότι είναι μία στις μας το να έχουμε διαφάνεια. Να είστε σίγουροι. Τι άλλο είπατε, τα κάτι μέλη, σωστή εφαρμογή, τι άλλο. Αυτή τη εβδομάδα είπαμε ότι θα ασχολούμεθα με το θέμα της προστασίας ιδιωτικού βίου και το και για τις διασυνορικές υποθέσεις. Έχουμε 73 τελικές αποφάσεις. Πέραν της ενεργοποίησης της διαδικασίας επίλυσης διαφόρων. Αυτές οι αποφάσεις εξεδόθησαν σε επίπεδο όπου υπήρχε αντιδικία, ελήφθησαν όλα υπόψη και καταλήξαμε στις 73 αποφάσεις. Εάν δεν είχαμε αυτό όλες τις εντυπωσιακές υποθέσεις, θα, ε, θα βλέπατε ότι κάμια φορά η μονοπεθεντική θηρίδα Μπορεί να σας φαίνεται ότι αργεί την περίοση αλλά τα κάνει ενδελεχώς όλα. Μα πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα. Παρακάτω. Ε, υλοποίηση της νομοθεσίας, κοινή δράση, τίποτα. PNR. Λάβατε την επιστολή μου, έτσι δεν είναι. Θέλετε να αναλάβουμε δράση άμεσα. Μα συμβαίνουμε στις διαπραγματεύσεις τα πάντα γύρω από το PNR. Και πιστεύουμε ότι μπορούν τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Και αν όχι καλύτερα, να έχουμε πιο ακριβή ρύθμιση στο μέλλον κοινέ δράσει εκτέλεση του νόμου. Αυτό είναι θέμα των εθνικών ευρωπαϊκών αρχών. Η εφαρμογή του νόμου είναι δική του αρμοδιότητα. Κοινή δράση. Σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό, προβλέπονται οι κοινέ δράσει μόνο εάν το προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για όλα τα κράτη. Αλλά συνεργαζόμαστε πολύ συχνά με όλους. με όλες τις εθνικές αρχές. Και όταν δεν προβλέπονται κοινέ δράσεις. Το DPC στην Ιρλανδία κάλεσε, ναι, κάλεσε ε, κάποιες εποπτικές αρχές. Τώρα, υποχρεωτική αποθήκευση δεδομένων. Για ξεκάθαρη τοποθέτηση. Ναι, είναι κρυστάλλινη θέση που έχω. Στο δε μέλλον θα τα πάμε ακόμα καλύτερα. Τώρα, η Ιρλανδική Υπηρεσία, εάν έχει προγραμματίσει σημαντικά πράγματα για το μέλλον, ναι, ισχύει αυτό και στα πλαίσια του IMI και σε αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε. Μέχρι τώρα όμως ε, αυτά τα σχέδια κειμένων δεν είναι στο σύστημα. Πριν εβδομάδα δόθηκε μία συνέντευξη όσον αφορά το τελικό κείμενο το οποίο θα δημοσιοποιηθεί αρχές του επομένου έτους. Πέρεκ. Σπούρεκ, Σπούρεκ, για την Πολωνία. Αυτούς τους 55 που είπατε ότι είναι ακόμα ε, έτοιμοι, όριμοι για το GDPR. Οι εθνικές αρχές βοηθούν, δίνουν κατευθυντήρες στις ε, εταιρείε, αλλά και σε οποιοδήποτε ενάγοντα για τα δικαιώματά του. Και στις μικρότερες εταιρείε. Βοηθάμε πολύ. Ονομοδοτούμε. Ρίστε μια ματιά στο πρόγραμμα εργασιών μας, ιδίως του 20. Τώρα να αφορά την ορθή εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη το κάνουν αυτό και η Κομισιόν επιβλέπει αν το κάνουν καλά. Και αν υπάρχει η ειδική νομοθεσία. Τώρα για την Ιταλία συνάδελφα, κυρία Κινίτση. Συγγνώμη, συγγνώμη, τα τελικά μου χολένα. Όσον αφορά τους ανηλίκους, στο πρόγραμμα εργασιών του 2020 έχουμε κάποιες κατευθυντήριες για τους ανήλικους και υπάρχει και κάποια ομάδα εργασίας με αυτό το θέμα. Και υπάρχει αυτό το δικαίωμα στη λύθη, το σβήσιμο δηλαδή, Έχουμε τέτοια ευθυντήρια γραμμή και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαβούλευσης. Πολύ ωραία. Τέλεια, τέλεια, λέει ο Πρόεδρος. Έκλεισε. Κλείδωσε. Κύριε Γέλνη, σας ευχαριστούμε. Α, πες κύριε Νεφέλτ. Σύντομη, σύντομη, γιατί έχουμε και άλλα δύο θεματάκια και κατόπιν 4,5 Θα είμαι σύντομη γιατί δεν είπατε τίποτα για το PNR, είπατε ότι συμβουλεύουμε κλπ. Τώρα όμως, τώρα όμως γίνεται μια παρέμβαση, είναι εξελίξη παραβίαση της νομοθεσίας. Γιατί δεν κάνετε τίποτα. Γέλνικ. Εκτός μικροφώνου. Ε, βέβαια. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι προβλέπετε. Ο πρώτος ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε το εναρκτήριο λάκτισμα σε σχέση με την επαφή με τον Ιόργανο, με την κυρία Γέλινεκ. Μας παρουσίασε την υπηρεσία της και επίσης το τι κατεύθυνε από τα πράγματα στο μέλλον και τώρα προχωρούμε. Καλώ όρισαν ναι, επίση οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας Γέλινεκ αλλά και του Ευρωπαίου του Δεδομένων τις καλύτερες αρχές μας του κ. και που είναι ο νέος επικεφαλής, ο νέος επόπτης. Περιμένουμε να έρθει η κυρία αυτή, με την περικυρία πρόκειται να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα. Σύντομος Και τώρα έχουμε τους επόμενους. Η επόμενη μισή ώρα θέλω κάθε ομιλητής να μιλήσει για 10 λεπτά, όχι περισσότερο, Οπότε έτσι να καταφέρουμε να στριμώξουμε λίγο χρόνο να μιλήσουν οι συνάδελφοι πριν έρθει η Επίτροπος Γιωχάνσον για τον διαρθρωμένο διάλογο. Μιλούμε τώρα για τα σημεία 4 και 5 που θα έχουν κοινή συζήτηση. Το θέμα ποιο είναι. Έχουμε την πρόταση κανονισμού τροποποιητικού του κανονισμού που διέπει το αίτιας. Βλέπω έχουμε τρεις προσκεκλισμένους. Τον ε, υποδιευθυντή της DG Home για το πρώτο και για το δεύτερο θέμα. Είναι ο κύριος υποδιευθυντής και κατόπιν είναι η, η κυρία Βάλβουλα. Εδώ την εξαριστερών μου. Α, έχουμε συναντηθεί στο πρωί Και παρακαλούμε να μας συνοψίσετε σε 10 λεπτά έκαστος και έτσι οι συνάδελφοι να μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις. Προτάσεις. Και όμως και το αναλυτικό σημείωμα, ούτω ώστε να δούμε πόσοι συνομοθέτες θα αποφασίζουν για, για αυτά τα δύο ε, ε, κείμενα του Ιανουαρίου του 19. Νιώδη Βαβουλά θα μας τα πει για το αιτίας. Uh, Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή. Να παρουσιάσουμε την πρόταση που πολύ τη γνωρίζετε. Είναι ένα από τα κατάλοιπα του, της προηγούμενης θητείας, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι ε, υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες ε, που βοηθήσατε να ε, προωθηθούν και τελικά να εγκριθούν πέρας αναβάθμισης της Frontex, ε, της τροποποίησης του συνορικού κώδικα του Σέγγεν για συστηματικούς ε, συνορικούς ελέγχους. Ε, μας βοηθήσατε λοιπόν πέραν αυτών και στην επικαιροποίηση και εξυγχρονισμό των διαφόρων ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών ως προς τον τύπο και ως προς την χρήση τους για τη διαχείριση των συνόρων. Επικαιροποιήθηκαν αυτά που ίσχυαν ήδη, το ΣΥΣ, το ΒΙΣ, το ΕΚΡΙΣ για τις υπηκός τρίτων χωρών, αλλά και νέα συστήματα δημιουργήθηκαν. Ένα από αυτά είναι το αντικείμενο της σημερινής ε, συνάντησης, το έτιας, ε, το μελλοντικό σύστημα προέγκρισης, που σημαίνει ότι θα έχουμε τον προτέρων πληροφορίες για όσους ε, ταξιδεύουν στην Ένωση χωρίς να έχουν θεώρηση διαβατήρια. Δηλαδή άτομα που δεν για το οποίο δεν είναι απαραίτητη η έκδοση θεωρησή. Είναι σημαντικό ε, για εμά ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε επαφή μαζί σα προ αυτό. Διότι ήδη εσεί είχατε θέσει τη νομική βάση και είχατε πει ότι είναι σημαντικό να οριστούν οι τρόποι και οι προποθέσει για να υπάρχει τη λειτουργικότητα μεταξύ αίτια και λοιπόν ε, πληροφορικών συστημάτων. Αυτή ήταν μια δέσμευση. Και η δεύτερη δέσμευση είναι ότι αν θέλουμε να λειτουργήσει το σύστημα αίτιας και να λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να μπορεί να έχετε και να ε, ρωτά, αν θέλετε, τα άλλα πληροφορικά συστήματα, άρα να έχει πρόσβαση σε όλα τα διαφορετικά συστήματα. Και το έκρης για επικοστριτών χωρών. Ο βασικός στόχος πρόταση ποιος είναι. Η εφαρμογή της αρχής ε, του privacy by design, δηλαδή ιδιωτικότητα μέσω σχεδιασμού. Έχουμε κάνει σχετικές προτάσεις βασιζόμενοι σε συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη. Υπό την έννοια ότι η πρόταση προσπαθεί να κωδικοποιήσει με ποιο τρόπο θα μπορεί να απευθύνεται αυτόματα στα διάφορα συστήματα πληροφοριών ε, που υπάρχουν το δηλαδή το Σέγγεν, ε, το ΒΙΣ και το ΕΚΡΙΣ, TCN, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για Επικός Τρίτων Χωρών. Επίσης, ε, θέλουμε να δούμε πώς θα μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες μετά από μία επισήμανση ότι κάτι εντόπισε το σύστημα. Και προβλέπεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο η διασύνδεση του συστήματος εισόδου-εξόδου και του συστήματος ε, πληροφοριών του Σέγγεν αντικαθεπτίζονται με το αίτιας και το σύστημα εισόδων-εξόδων. Κάθε φορά που κάποιος φτάνει στα σύνορα της Ένωσης, έχοντας καταθέσει το αίτημα προέγκρισης αίτιας, ε, τα δεδομένα αυτά θα ελέγχονται με το σύστημα εισόδου-εξόδου που είναι η βάση, το σημείο αναφοράς, που σε πραγματικό χρόνο θα επικαιροποιεί τις προφορές για αυτούς που μπαίνουν ή φεύγουν από την Ένωση. Ένα είδος μητρώου για να βλέπουμε κατά πόσον κάποιος έχει περβεί τον χρόνο διαμονής, παραμονής που τα τρεπόταν. Πολλές ήταν οι ερωτήσεις ε, που μας θέσατε. Δεν θεωρήσαμε ότι χρειάζεται μία πλήρης μελέτη αντικτύπου και γιατί κάποιες φορές ε, έχουμε ως υπεργολάβου εσάς στο Κοινοβουλίο, αλλά θα τα δούμε και αυτά, αλλά γιατί και η νομική βάση το έτσι ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος προς το τι έπρεπε να γίνει. Δεν έχουμε περιθώρια λιγμών. Άρα ουσιαστικά εφαρμόζουμε τις προηγούμενες αποφάσεις των συνομοθετών. Όχι δηλαδή μελέτη αντικτύπου, αλλά ένα επεξηματικό σημείο αναλυτικό με πρόταση και με βάση τις ερωτήσεις που μας ε, στείλατε, ε, εκπονήσαμε και ένα αναλυτικό σημείωμα ξεχωριστό. Χρειαζόμαστε ε, ασφάλεια δικαίου προς το ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα και γιατί θα χρησιμοποιούνται. Δεν θέλουμε να υπάρξει κάποια παρέκκληση από όλο το πλαίσιο που αφορά τη διαλειτουργικότητα και το οποίο έχουν εγκρίνει οι συνομοθέτες. Υπάρχουν πολλές αρχές, υπάρχουν κριτήρια τα οποία είναι σωματωμένα στις νομικές βάσεις των διαφόρων συστημάτων που και αυτά πρέπει να τηρηθούν. Πρόκειται για, αν θέλετε, μια μηχανική μετάφραση του τι είναι απαραίτητο ώστε το αίτιας να μπορεί να ρωτή ε, ρωτήσει όλα τα συστήματα και στα νέα και στα ε, και παλιά. Ο Καινούργιο όπως το έκρισε για τους 23 των χωρών. Μας βοηθήσετε πάρα πολύ και τηρήσετε και το χρόνο σας. Ευχαριστώ κύριε Βαβουλά, έχετε εσείς τώρα το λόγο. Βάβουλα, Βαβουλά, πώς λέγεστε. Βάβουλα λέγομαι. Kind invitation. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ευγενική πρόσκληση και η, εταιρεία, η υπηρεσία έρευνας κοινοβουλίου ανέλαβε αυτή την ε, μελέτη. Ελπίζω μέσα σε 10-15 λεπτά όσο διαρκέσει δηλαδή η παρουσίασή μου, ε, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω ποια τα βασικά πορίσματα. Και πρώτα απ' να σας πω, πρόκειται για στοχευμένη μελέτη, ε, δηλαδή ήταν δύο τα βασικά ερωτήματα τα οποία αναλύσαμε. Δεύτερον, ποια ήταν η μεθοδολογική προσέγγιση, ποια είναι τα βασικά πορίσματα σας το κάθε ερώτημα και θα τελειώσω κάνοντας κάποιες συστάσεις και κατάλληλες κάποια συμπεράσματα. Δεν έχω βέβαια τη δυνατότητα να σας εξηγήσω 30.000 λέξεις ανάλυση, ελπίζω όμως η ανάγνωση της μελέτης να σας ικανοποιήσει. Για τα δύο ερωτήματα, ποια ήταν. Πρώτον, σε ποιο βαθμό οι δέσμοι μέτρων της Κομισιόν επεκτείνει το πεδίο σε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Γλυφαπίνικου Μητρώου για του των χωρών και κατά πόσον η επέκταση αυτή δημιουργεί κάποιο πρόβλημα ή πρόκληση σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά και την προστασία τη ιδιωτική σφαίρα. Το δεύτερο για τη δέσμη μέτρων ερώτημα ήταν αν οι κανόνε για την αυτόματη εξεργασία ετοιμάτων μέσω του έτες με διασταύρωση όλων των άλλων συστημάτων πληροφοριών, αν και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα και προκλήσεις ε, για τους τομείς που προανέφερα, προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα. Μεθοδολογία. Ήταν πάρα πολύ σύντομο το χρονοδιάγραμμα, ε, από τα τέλη Οκτωβρίου έως την προηγούμενη Παρασκευή που δώσαμε στη δημοσιότητα το σχέδιο της τελικής έκθεσης. Αυτό ήταν ο χρόνος, πολύ περιορισμένος. Και επομένως περιορισμένο και η μέθοδος. Βασιστήκαμε στην δοκιμαστική έρευνα, αλλά με τη γάμα Δελτα Home, η ο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Επόπτη, κάναμε συνεντεύξεις σε αυτούς ε, και τους ενημερώσαμε για τα βασικά προκατρακτικά πορίσματα. Ένας άλλος περιορισμός πέραν του χρόνου ήταν οι διαθέσιμες πληροφορίες. Βασιστήκαμε στις ε, δημοσία διαθέσιμες πληροφορίες και επειδή αυτό το πακέτο της Κομισιόν είναι έτσι διαδρομένο ώστε μόνο τις τροπολογίες περιλαμβάνει. Εγώ έπρεπε να καταρτήσω ένα πίνακα με όλες τις αλλαγές σε σύγκριση με το τρέχον νομικό πλαίσιο. Αυτό το βλέπετε στο τέλος της μελέτης. Καταλήγοντας, επειδή είναι μελέτη για θεμελιώδη δικαιώματα αυτή, έγινε εκτίμηση με βάση την ομολογία των δύο Ευρωπαϊκών Δικαστήριων, λαμβάνοντας υπόψη βασικές αρχές προστασίας δεδομένων. Πρώτο ερώτημα, λοιπόν, για την επέκταση του πεδίου εφαρμογή με το έκρηστη Επεκτείνει το πεδίο πέραν των συμπεφωνημένων ε, στον κανονισμό έκρηση για υπηκός τρίτων χωρών του Ιουνίου του 2019. Στον κανονισμό αίτιας πράγματι έχουμε την Ατολική Σκέψη 18 που λέει ότι αν θεσπιστεί τέτοιο σύστημα έκρηση για επικό τρίτων χωρών θα πρέπει να μπορεί το αίτιας να έχει πρόσβαση, αλλά κατά την άποψή μου δεν είναι επαρκή νομική βάση η τολική σκέψη, γιατί δεν έχουν οι τολικές σκέψεις δεσμευτικό χαρακτήρα. Είναι μόνο ερμηνευτικό ο χαρακτήρα του. άρα δεν είναι επαρκή. Τώρα, για την επέκταση, ε, δεν υπήρξε ο δέον έλεγχο, έλεγχος, για την ε, έγκριση του κανονισμού που δεν βασίστηκε σε μελέτη αντικτύπου, αλλά σε μελέτη σκοπιμότητας, αλλά σε ό,τι αφορά τον κανονισμό έκρησης και το πακέτο αυτό, πάλι ε, υπάρχει κενό σε ό,τι αφορά τη μελέτη αντικτύπου, τριπλό δηλαδή κενό. Έχουμε τα 7 και 9 του χάρτη, δικαίωμα στη ιδιωτικότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων. Εδώ μιλάμε για μια σοβαρή παρέμβαση. Μιλάμε για μια βάση δεδομένου έκρηση της ΣΥΕΝΗ, η οποία εγκρίθηκε με βάση μια νομική βάση για την επιβολή της νομοθεσίας, ενώ τώρα θα χρησιμοποιηθεί για στόχους, σκοπούς ε, διαχείρισης συνόρων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η παρέμβαση, ότι δηλαδή υπάρχουν νέε μορφέ επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νέε αρχέ που τα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα στο έκθεση και σε ό,τι αφορά την σκοπιά αυτή τη προστασία δεδομένων, αυτή η επέκταση δύσκολα συμφιλώνεται και με την αρχή του ε, περιορισμού του πεδίου εφαρμογή που είναι βασικό στοιχείο τη σχετική νομοθεσία. Δηλαδή δεν είναι σαφή τα όρια μεταξύ ε, του νόμου για, νομοθεσία, για τη μετανάστευση, για την προστασία συνόρων, ε, για την προστασία δεδομένων. Δηλαδή άλλη σκοποί για τους οποίους αρχικά δεν υπήρχε πρόβλεψη. Αυτό που έπρεπε λοιπόν να εξολογήσουμε κατ' αν η αρχή της αναγκαιότητας αναλογικότητας του άρθρου 52 του χάρτη, αν αυτές γίνονται σεβαστές και αιτιολογούν την επέκτηση που παιδιφαρμολισμού με το έκριση Αποτέλεσμα. Θετικό είναι ότι το έκριση όχι μπορεί να θεωρηθεί θετικό γιατί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι αρχές ε, μετανάστευση ή έλεγχου συνόρων. Αυτό επιτρέπει εθνική νομοθεσία αλλά και με την προσέγγιση των ΗΠΑ είναι συμβατό όταν χρησιμοποιούν ε, ε, το ΕΣΤΑ, το αντίστοιχο αυτό σύστημα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία ποινικού μητρώου αλλά δεν συνάδει με την προσέγγιση ε, του Αυστριαλιανού ΕΤΑ, που είναι το αντίστοιχο ευρωπαϊκό αίτιας, ε, όπου πρόσβαση δίνεται μόνο σε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις, όταν έχουμε ένα alert. Τώρα, το πακέτο κάνει μια διάκριση μεταξύ τρομοκρατικών αδικημάτων και σοβαρών αξιόπινων πράξεων. Καλό αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι αν είναι αναγκαίο τελικά ε, να υπάρχει πρόσβαση στο έκρηση της ΙΕΝ το ΣΥΣ. Από ό,τι ξέρω, αποθηκεύει ήδη ε, κάποια σήματα, κάποια alerts για 20 χρονών. Άρα αυτό θα σημάνει άλλη μεταξύ του δεύτερου ΣΥΣ και του έκρηση της ΙΕΝ. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα υπάρξει αυτή η επικάλυψη. Γιατί. Διότι το δεύτερο ΣΥΣ ε, στον κανονισμό το αναφέρεται ότι η καταδίκη για τρομοκρατικά δικήματα πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρίζεται στο έκρηστη ΣΥΕΝ, αλλά σε ό,τι αφορά άλλε αξιόπινε πράξει δεν είναι αυτό δυνατό. Επομένω, δεν ξέρουμε ακριβώ σε ποιο βαθμό θα υπάρξει αυτή η αλληλεπικάλυψη. Αλλά όλα οι σοβαρέ υποθέσει πιστεύουμε θα μπουν στο δεύτερο ΣΥΣ. Και δεν υπάρχει κάποια έδειξη ότι το ε, σύστημα με τι προειδοποιήσει, με τα alert δεν επαρκεί. Επίση, ό,τι αφορά την επισήμανση, το flagging, ότι πρέπει να υπάρξει κάποια ε, διάκριση για τους ε, πολίτες διπλής υπηκότητας που μπορούν να απολαμβάνουν δικαιωμάτων ελεύθερης διακίνησης και μπορεί να μην χρειάζονται όλα αυτά. Περνάω στο δεύτερο ερώτημα. Οι κανόνε για την αυτόματη επεξεργασία νομίζω είναι ε, άρτη και ισορροπημένοι. Υπάρχουν κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδε ε, ώστε η κεντρική μονάδα του αίτιας και οι εθνικές μονάδες του αίτιας να μην έχουν πρόσβαση σε μητρώα ε, ε, κατά τρόπο που δεν θα είναι αναγκαίος. Πώς θα το αξιολογούσαμε αυτό όμως. Γι' αυτό χρησιμοποίησα ε, τα guidelines από την γνωμοδότηση 1.15 στο τέλος τα, τα στοιχεία PNR και βλέπω στην ανάλυση μου ότι μπορεί μεν να είναι ισορροπημένοι οι κανόνες. Θα υπάρξουν όμως κάποια ζητήματα. Παραδείγματο χάρη πρόβλημα ποιότητα, Το βλέπουμε αυτό δυστυχώς σε όλα τα συστήματα πληροφοριών, τυπογραφικά, σφάλματα κτλ. Γίνονται προσπάθειες διόρθωσης, αλλά όσο ε, πιο πολύ ε, τη συμβουλεύεται κάποιο σε αυτή τη νομική βάση, θα υπάρχουν αυτά τα λάθο ε, hit και άλλες ε, παρατυπίες και ανομαλίε. Υπάρχει ένα πρόβλημα αποθήκευσης κάποιων λιμάτων που δεν γίνεται με νόμιμο τρόπο. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες καταγγελίες. Για το ΒΙΣ τα δεδομένα μπορεί να μην είναι πάντοτε ε, συναφή, επειδή έχουν τελείως διαφορετικό πεδίο εφαρμογή στο ΒΙΣ από το ΣΥΣ. Άλλοι κανόνες, διασταύρωση ε, κάποιων ελέγχων, νομίζω ότι είναι σωστό. Κανόνες για την άμεση ε, ε, είσοδο δεδομένων από το αίτια ε, στο σύστημα εσόδων-εξόδων δεν είναι κάτι που αιτιολογείται. Αλλά από τη δική μου τη μελέτη προκύπτει ότι όλα αυτά δεν είναι τεχνικέ προσαρμογέ. Έπρεπε να έχει γίνει μελέτη αντικτύπου σε κάποιο χρονικό σημείο, γιατί έχουμε αυτό το τριπλό κενό που προανέφερα. Ούτε αιτιολογείται και είναι και πλήρω αναγκαίο η επέκταση που θα καλύψει το έκρηστη σένα, αλλά οι άλλοι κανόνε ε, έχουν καταρριστεί με προσοχή Άρα, όπω θα δείτε στη μελέτη, υπάρχουν και κάποιες συστάσεις για το πώ περαιτέρω μπορούμε να διευκρινίσουμε και να αποκρισταλώσουμε τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα και στις των δεδομένων. Βαβούλα, now. Ευχαριστούμε κυρία Βάβουλα. Θυμηθείτε ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε έξω την Επίτροπο να μας περιμένει. Πρώτη φορά έρχεται η Επίτροπο στην Επιτροπή μας. Δεν θα πρέπει να ε, τη στήσουμε θέλει να μας παρουσιάσει το πρόγραμμά της για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μας έχει υποσχεθεί να το φέρει και να το παρουσιάσει το πρώτο τρίμηνο του 2020. Να ακούσουμε λοιπόν αυτούς που ενέχονται με τις εκθέσεις αυτές άμεσα πρώτα τον εισηγητή, τον κύριο Λέναρς και μετά του Σκιώδης, αλλά παρακαλώ ε, αναφερθείτε επιγραμματικά μόνο στα πιο σημαντικά. Μα είναι τόσο πολλά τα σημαντικά. 12 λεπτά έχουμε τώρα, τι να κάνω. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και θα τα ξαναδούμε, θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε. Χαίρομαι πολύ που μπορούμε επιτέλους να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Είναι οι συνέπειες ε, ε, όσων αποφασίσαμε την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο. Συμφωνώ με την κυρία Νιώβη Βάβουλα ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μελέτη αντικτύπου από την αρχή, ιδιαίτερα για το ETIAS δεν είχε στην αρχή χάρη στη δική σας σκληρή δουλειά. Τώρα αυτό είναι γεγονός και μπορούμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε και χαίρομαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα αίτιας που να λειτουργεί σωστά, θα πρέπει αυτές οι, τροπολογίες, ε, οι τροποποίησεις να περάσουν. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσατε να μας απαντήσετε και για τη μελέτη αντικτύπου ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πρόβλημα λειτουργίας που ανέφερε η κυρία Βάβουλα. Και δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν έχετε βάλει και ειδοποίηση για τις επιστροφές. Όταν κάποιος επιστρέφει μετά από απόφαση επιστροφής, διαγράφεται αυτή η ειδοποίηση αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη διαδικασία και άρθρο 8, αν κάτι πάει στραβά, να μην κρατείτε στα σύνορα κάποιος για 12 ώρες, ενώ είναι ακόμα στη διαδικασία διαβούλευση, ειδικά για το αίτιας, Όταν κάποιο έχει φύγει ε, και έχει παραμείνει ακόμα η ειδοποίηση επιστροφής, δεν έχει διαγραφεί και φαίνεται ότι παραμένει στην Ένωση, υπάρχουν προβλήματα. Πάνε και τους κρατάνε στα σύνορα 12 ώρες. Ε, και για το ΒΙΣ, το σύστημα ενημέρωσης για τις θεωρήσεις, εκεί πώς θα εξασφαλίσετε ότι υπάρχει ε, σωστή εφαρμογή για την έρευνα σχετικά με τη μελέτη που εξεπλάγει λίγο όταν είπατε για την επέκταση του ETSTCN. Απέφυγε τον έλεγχο και πέρασε κάτω από τα ραντάρ και εγκρίθηκε χωρίς να ε, υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Μα είναι στη διαδικασία συναπόφασης και προσέχουμε πάρα πολύ και τα άρθρα και ε, τις τροπολογίες και τις αιτιολογικές σκέψεις και φροντίζουμε να υπάρχει πάντα η απαραίτητη πλειοψηφία για να περνάνε και στο Συμβούλιο τα ίδια. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα ότι διέφυγε του κοινοβουλευτικού ελέγχου και το περάσανε στη ζούλα. Όπως είπατε κι εσείς, το αίτια TCN στήθηκε ακριβώς για να βοηθάει τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται τα σύνορα, τη μετανάστευση, τις θεωρήσεις κτλ. Θα με ενδιαφέρε η απάντησή σας. Και επίσης, το έκρις TCN, όχι αίτιας, έκρις, συγγνώμη, και οι ειδοποιήσεις για το άρθρο 24 ε, στο SIS δεν αντιστοιχούν πάντα σε ε, καταδικασθέντες ε, πολίτες τρίτων χωρών. Αν δεν το συμπεριλάβετε, θα υπάρχουν ελλείψεις και κενά. Για να είναι πλήρες το σύστημα θα πρέπει να συμπεριλάβει. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια άρνηση ή ειδοποίηση σε ό,τι αφορά την είσοδο, ε, αν δεν αναφέρεται καταδίκη καταδίκη, κάτι λείπει. Εν πάση περιπτώσει, δεν επεκτείνομαι. Ε, με πολύ μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ με όλου τους συναδέλφου. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας. Και τώρα πάμε στους κοιόδη. Με τη σειρά. Πρώτος, ο κύριος Μωράε από τους Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπω είπε ο κύριος Λέναρς, ε, αυτά ήταν τα σημαντικότερα και με κάλυψε. Αύριο θα συνεδριάσουμε σκιώδε και θα μπορέσουμε να το δούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το βασικό πολιτικό ζήτημα για μένα αυτή τη στιγμή είναι το εξή. Για ποιο λόγο ζητήσαμε αυτή τη μελέτη αντικτύπου. Διότι αναπόφευκτα στη μελέτη EPRS της δική μα ε, υπηρεσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπήρξε λεπτομερή ε, εστίαση στα θεμελιώδη δικαιώματα, στην προστασία πολιτικών δεδομένων και σε άλλα. Ε, είναι πολύ μεγάλο το θέμα και δεν θα μπορούσε να το καλύψει η δική μας μελέτη. Αλλά και, όπως είπε και ο κύριος Λέναρς, υπάρχουν πολλά θέματα που είναι σημαντικά και θα εξετάσουν οι σκιώδεις, αλλά δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τα καλύψουμε όλα. Έχουμε μια μελέτη από το EPRS, που δεν είναι η βασική μελέτη, ε, Υπάρχουν λοιπόν κάποια κενά στην εφαρμογή. Και το έκρις TCN ε, τώρα παρατείνεται, επεκτείνεται αλλά είπατε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην προστασία προσωπικών δεδομένων κτλ. Το έκρης TCN θα χρησιμοποιηθεί για αλότριους σκοπούς από εκείνους που είχαν ε, σχεδιαστεί. Θα υπάρχει κίνδυνος δηλαδή αποκλίνουσας εφαρμογής. Δεδομένων λοιπόν αυτών των ευρημάτων σας, εν μέρη απαντήσατε στην παρουσίασή σας, αλλά τα βασικά ερωτήματα είναι εάν συνάδουν με τον κανονισμό αίτιας τα όσα ισχύουν αυτό τον καιρό, αν χρειάζονται αλλαγές τεχνικές και τα συμπεράσματα της μελέτης σας έδειξαν. Το πεδίο εφαρμογή επεκτάθηκε. Αυτό τώρα σημαίνει επέμβαση στα ανθρώπινα ε, δικαιώματα, στα θεμελιώδη και στην ιδιωτικότητα και στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Και οι τροπολογίες για την τελική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επεμβαίνουν στην ιδιωτικότητα και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Είναι βασικά αυτά τα σημεία, θα τα συζητήσουμε αύριο στην εδρία των σχεδών. Αυτό όμως που ήθελα να επαναλάβω και να τονίσω είναι ότι καλό θα ήταν να αρχίσουμε, καλύτερο μάλλον, ε, από μια ευρεία μελέτη αντικτύπου. Αναφέρθηκε ο κύριος Λέναρ αυτό. Θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στην επιβολή του νόμου και στο δίκαιο ασύλου ή μετανάστευσης δεν θα πρέπει ε, για να λύσουμε ένα πρόβλημα να κοιτάμε ε, λάθος βάσεις δεδομένων και να έχουμε πρόσβαση σε λάθος προσωπικά δεδομένα. Στόχος είναι να, να τρέχουμε στις σωστές βάσεις δεδομένων και να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που μας χρειάζονται και όχι να εισβάλλουμε στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Το Renew, σύντομα παρακαλώ όσο μπορείτε. Όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί τα είπαν οι συνάδελφοι που ήθελα να πω, όσο το πλήστο. Όταν το διάβασα και εγώ θεώρησα ότι τίποτα απλό δεν υπάρχει σε αυτές τις ε, τροποποίησεις. Είναι θέματα ουσίας που είπε και ο κύριος Μωράς. Αυτό είναι η ουσία της ε, πρότασης, η διαλειτουργικότητα, πώς γίνεται, ποιες είναι οι επιπτώσεις και για το τι προκύπτει, αλλά και καθ' αυτή η διαλειτουργικότητα. Καλά πάντως αύριο θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Αλλά έχω και στους δύο προσκεκλημένους αυτό το function grid. Αυτό το κίνδυνο αποκλίνουσας εφαρμογής. Γιατί επιφυλάσσουμε όσον αφορά αυτά τα επιχειρήματα της μελέτης, όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει νομική βάση για ασφάλεια. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Καλά, μην προδικάσω το που θα καταλήξουμε. Θέλω να μου πείτε τη σκέψη σας. Και επιτροπή να μου πει, υπάρχει ή δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Κύριο Λέναρτ, τι μα είπε. Μα είπε για το κατά πόσον υπάρχει επικάλυψη του αιτιάς με το ΒΙΣ σε σχέση με κάποιους που έχουν καταδικαστεί. Το SIS δεν καλύπτει ε, αυτό το ενδεχόμενο, ούτε το έκρισε Και επίσης μας είπατε και για τα δεδομένα του VIS για την αναζήτηση των δεδομένων και είπατε δεν χρειάζεται να υπάρχει αναζήτηση από τη μία πλατφόρμα στην άλλη. Μα ένα σωρό χώρες πρόσφατα έχουν κόψει τις βίζες και άρα τώρα θα χρησιμοποιείτε το αίτιος. Στο παρελθόν όμως χρησιμοποιείται το, το VIS για να ταξιδέψει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις θεωρήσεις που υπήρχαν είναι εδώ πέρα θέματα ε, διαχείρισης ε, έλεγχων συνόρων, ασφάλειας. Γι' αυτό πέστε μου τη γνώμη σας. Αυτά. Και εσείς και εσείς κύριε από τους Πρασίνους, ε, πέστε μας. Μπράια. Πολύ θετική η μελέτη σας που μας εξηγεί τα όρια μεταξύ δικαίου μετανάστευσης και εφαρμογής του νόμου. Και εμείς από την αρχή έχουμε επικρίνει το αίτιας Χρειάζεται καλύτερη τεκμηρίωση για να κάνει κανείς ε, τέτοιες ε, κάποια νομοθεσία. Να μην καταλήγουμε σε διακρίσεις. Πολλά ε, που ήθελα να πω τα είπαν οι συνάδελφοι, οπότε δεν ρωτάω παραπάνω και παίρνω να ακούσω τις απαντήσεις. Ο Πρόεδρος. Και τώρα. Ο κύριος Λάς Πάτρικ Μπέρκ είναι εδώ. Όχι. ECR, ούτε από το ECR έχουμε σκιώδηση, γιατί η Σοφή Πελετιέ της Γκουέ όμως είναι εδώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι αρκετά σύντομη, γιατί έχω βραχνιάσει όλες, δεν ξέρω να με ακούτε, ελπίζω να με ακούτε. Για το έκρης και το αίτιας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές στα κράτη-μέλη ανάλογα με τις κυρώσεις, με τις αξιόπινες πράξεις και για το πώς εγγράφονται στα Μητρώα ε, οι εγκληματίες γιατί δεν είναι εναρμονισμένα τα ποινικά συστήματα. Παραμένω εγώ πολύ προσιλωμένη στο γεγονός ότι ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει πραγματική μελέτη αντικτύπου γιατί κατά την άποψή μου αυτά τα θέματα δεν είναι αμυγός τεχνικά, είναι και πολιτικά και αν αυτή η μελέτη αντικτύπου θα πρέπει να επικεντρωθεί σε κάτι τόσο ειδικό αυτό είναι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ για αυτά. Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Πελτιέ. Προτείνω τώρα επειδή έχουμε και άλλο ραντεβού αμέσως μετά, στις 9 Ιανουαρίου, όπου ο εισηγητής θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής της και του, θα παρακαλούσαν να σταματήσει η συζήτηση ε, στους ε, σκιώδεις και να απαντήσουν σύντομα οι ε, ομιλητές μας, για να έρθει και επίτροπος. η κυρία Γιώχανσον, η οποία ήδη περιμένει, ε, μάλλον έχει ήδη μπει στην αίθουσα. Ε, καλωσορίσατε και ε, λίγα λεπτά υπομονή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σονιντή, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί είναι εδώ η Επίτροπός μου και δεν θέλω να την αφήσω να περιμένει. Σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως, για να επανέλθω σε αυτό. Δεν είναι ε, σωστό για το περιεχόμενο της πρότασης, αν το χαρακτηρίζουμε το θέμα τεχνικό. Είναι προσωπικά δεδομένα και πώς ε, ε, έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Δεν είναι απλό θέμα, αλλά έχει συνέπειες. Όπως είπε και ο εισηγητής, ουσιαστικά στην πράξη μεταφράζει κάποιες αποφάσεις που έχουν λάβει οι συνομοθέτες. κατέρωθεν. Και εδώ έχουμε μια μικρή διάσταση απόψεων σε σχέση με το πόρισμα της ε, μελέτης και ζητώ συγγνώμη που δεν την έχω διαβάσει ακόμα, αλλά αυτό η αιτιολογική σκέψη για την απόφαση αίτιας είναι πολύ σαφής. Ε, ε, πολύ σωστά είπατε τι είναι αιτιολογική σκέψη. Περιγράφει, εξηγεί, ερμηνεύει το κείμενο, αλλά κάποιος ορίζει το πεδίο εφαρμογής που περιγράφεται εκεί. Για το έκρις, για όσους έχετε εργαστεί στο έκρις της ΙΕΝ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι εσείς ε, ε, τροποποίησατε κάποια χαρακτηριστικά της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έκρης της ΙΕΝ, ακριβώς διότι έδινε πρόσβαση στο αίτιας. Ας πούμε επιλέξατε και δικαιολογήσατε ε, τι πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται και κρατούνται και τηρούνται εκεί στο σύστημα έκρης TCN ακριβώς για να ε, είναι ε, διαθέσιμο και να χρησιμοποιείται στα πλαίσια της προέγκρισης του αίτιας. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν νομίζω ότι είμαστε σε πολύ γερό έδαφος. Ένα δεύτερο. Το θέμα δεν είναι τόσο πολύ αν έχει αλλάξει ο σκοπός ή όχι. Όχι, δεν έχει αλλάξει. Παραμένουμε πολύ στη διαχείριση των συνόρων. Και συζητούμε πώς ελέγχουμε ε, τα σύνορα, πώς οργανώνονται αυτοί οι έλεγχοι στα σύνορα και τι εργαλεία χρησιμοποιούμε για να διεξάγονται οι έλεγχοι αυτοί. Αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα. question... Το σημαντικό λοιπόν και το κύριο ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο ορίζεται η αρχή της αναγκαιότητας. Δηλαδή αποκαλύπτουμε και χρησιμοποιούμε τις προφορίες που είναι απολύτως απαραίτητοι για τους συνοριακούς ελέγχους. Και έχουμε και πλήρη ε, σαφήνεια ε, στο μυαλό μας για την αλληλουχία των γεγονότων. Πολύ σημαντική διάκριση. Τι γίνεται αυτόματα ας πούμε ε, με μια σημείωση flag, ναι ή όχι, είναι γνωστό αυτό το πρόσωπο ε, στις αρχές ε, σε κάποιο σύστημα πληροφοριών που υπάρχει για κάποιο λόγο και μετά υπάρχει πολύ συγκεκριμένη διαδικασία κωδικοποιημένη για τον τρόπο με τον οποίο έχει κανείς πρόσβαση και για ποιους λόγους και αυτή είναι πολύ περιορισμένη. Και για το VIS ε, θα ε, βεβαιώσουμε στον επόμενο τριμερή διάλογο που γίνεται αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη συγκεκριμένα, ότι θα υπάρχει πλήρη συμμόρφωση. Ε, υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη για όσους έχουν διπλή επικότητα, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μια ειδική κατηγορία. Based Αλλά με βάση τα σχόλια που δεχτήκαμε, που λάβαμε και χάρη στην προθυμία του εισηγητή να αρχίσει πολύ γρήγορα τη δουλειά, τώρα είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας και περιμένουμε ε, ε, εναγωνίως να αρχίσουμε τη συζήτηση σε βάθος. Η κυρία Βάβουλα, ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Πάρα πολύ σύντομα για το ΣΥΣ, Σύστημα Πληροφοριών Σέγγεν. Λέω στη μελέτη μου ότι είναι άγνωστη η επικάλυψη, ο βαθμός της επικάλυψης, αλλά ο στόχος αυτών των ειδοποιήσεων είναι ακριβώς να αποφευθεί η είσοδο συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών ε, τρίτων χωρών. Αν θεωρούν κάποια κράτη-μέλη ότι δεν θα πρέπει να μπει στο Σέγγεν ε, ένας πολίτης τρίτης χώρας που έχει καταδικαστεί, θα υπάρχει ειδοποίηση, σήμα, alert. Και δεν υπάρχει τίποτα πουθενά που να λέει ότι τα κράτη-μέλη ε, ε, δεν ε, εισάγουν στο σύστημα με ικανοποιητικό τρόπο αυτά τα σήματα της ειδοποίησης. Μπορεί να μην είναι ακόμα πλήρες το σύστημα, αλλά θα είναι αρκετά επαρκές, έτσι ώστε να μην δικαιολογείται η επέκταση του συστήματος έκρησης TCN. Κατανοώ ότι η αιτιολογική σκέψη θεωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμευτική, αλλά κατά την άποψή μου αν δεν έχει γίνει σωστή μελέτη αντικτύπου ε, σε πολλές περιπτώσεις για ένα ζήτημα, αυτό σημαίνει ότι έχει διαφύγει το ελέγχο και έχει περάσει κάτω από το ραντάρ. Και πρόκειται ε, για βάσεις δεδομένων που έχουν ε, ποινική προέλευση και ε, σοφρονιστική επιβολή του νόμου. Και δεν μπορεί να αναμειγνύονται όλα στο μέλλον, στο ίδιο πεδίο. Και σε κάποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρόταση κινδυνεύει να οδηγήσει σε αυτή την ανάμειξη που έχει ήδη γίνει και πρέπει να σταματήσει. Σε ό,τι αφορά το VIS και τα λοιπά, σας παραπέμπω στη μελέτη ε, όπου υπάρχει ένα ειδικό σημείο, μια ειδική σημείωση για τους πολίτες με διπλή υπηκοότητα, ε, όπου η μία χώρα είναι στη μαύρη λίστα και άλλη στην άσπρη. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα προς το παρόν. Η μελέτη είναι στη διάθεση όλων σας και εγώ φυσικά στη διάθεσή σας για τις μελλοντικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για τη συντομία για να μην καθυστερήσει πάρα πολύ η επόμενη συζήτησή μας με την Επίτροπο. Κύριε Τουντοράτσε. ευχαριστώ. Ε, συγγνώμη. Ε, καθυστέρησα και δεν πρόλαβα να διαβάσω τη μελέτη. Τι περιθώριο χρόνο έχουμε. Μπορείτε να μας απαντήσετε γραπτώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σημεία της μελέτης ως δική σας απάντηση, επόκριση στη μελέτη για να κατανοήσουμε και όλα τα επιχειρήματα από όλες τις πλευρές. Καλωσορίζουμε θερμά την κυρία Γιώχανσον, Επίτροπο Ορμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις. Ελάτε παρακαλώ. Η πρώτη φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας in charge Ως επίτροπος πλέον ε, έχει αναλάβει τα καθήκοντά της και το χαρτοφυλάκιο αυτό. Thank you all. Thank you all. Now, as I said, we have one hour. Όπως σας είπα, έχουμε μία ώρα. Um, yes, one hour, 45 minutes. Και 45 λεπτά. Έτσι δεν είναι. But it'll be one hour 20. According to the, uh, to the uh, time... Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε προβλέψει, γιατί έχουμε και ψηφοφορία. Και ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα με τις ψηφορίες. Έρχεται ο κόσμος τρέχοντας, ακριβώς την ώρα που έχουμε προβλέψει για να ψηφίσει. Λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε για πρώτη φορά την Επίτροπο κυρία Ήλβα Γιώχανσον, αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις. έχει το άσυλο, τη μετανάστευση, την εσωτερική ασφάλεια, το μέλλον του Σέγγεν. Είναι θέματα πάρα πολύ προσφυλή σε μας. Και μεταξύ αυτών και το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Μέγα θέμα. Ήδη έχει αρχίσει περιοδία στις πρωτεύουσες μαζί με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Σχοινά Τις τελευταίες μέρες πήγατε στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Την καλωσορίζουμε και περιμένουμε να ακούσουμε την παρουσίασή της στο πλαίσιο του λεγόμενου διερθρωμένου διαλόγου που σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την κυρία Γιωχάνσον για τα θέματα της δικής της αρμοδιότητας. Θα ήθελα επίσης, κυρία Γιώχανσον, να σας προσκαλέσω ρητά να έρθετε στο διάλογο που θα κάνουμε, διάλογο ασφαλείας μετά τις διακοπές με τον Τζούλιαν Κίνγκ που είχε αυτή την αρμοδιότητα στο παρελθόν. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και μαζί σας αυτό το διαρθωμένο διάλογο για τη στρατηγική εσωτερική ασφάλεια. Και αυτό είναι μια ευκαιρία και για τα δύο θεσμικά μας όργανα να έχουμε μια εις βάθος ανταλλαγή απόψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αρχίζουμε λοιπόν, θα πάρετε το λόγο για ένα τέταρτο. Ήδη σηκώνονται κάρτες. Μια μισή ώρα έχουμε, όχι παραπάνω. Ε, να το έχετε υπόψη σας, παρακαλώ να κάνετε τις ερωτήσεις σας όσο γίνεται πιο σύντομα και πιο άμεσα. Καλώς ορίστε και πάλι κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Θα ήθελα να μοιραστούμε τις απόψεις σου για το χαρτοφυλάκιό μου και τι προτίθεμαι να κάνω, αλλά ήρθα κυρίως για να ακούσω τις δικές σας προτάσεις και τις δικές σας απόψεις και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την εσωτερική ασφάλεια. I think the issue of Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας έχει να κάνει με τη συνοχή σε μια κοινωνία. Έχουμε δει το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα να αυξάνεται σημαντικά. Έχουμε απειλές από τρομοκρατικές ομάδες. Βλέπουμε τεράστια αύξηση της χρήσης ναρκωτικών που συνήθως έτσι το οργανωμένο έγκλημα ε, χρηματοδοτεί τη δράση του, ε, αυξάνονται και πληθύνονται πολύ γρήγορα με νέα επιχειρηματικά μοντέλα για να το πω. Ε, είναι πραγματικά εγκληματίες και δρούν διασυνοριακά οι περισσότερες αυτές ομάδες. Εκεί πραγματικά υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία εάν το αντιμετωπίσουμε το θέμα ευρωπαϊκά. Για μένα ακριβώς αυτό έχει να κάνει με την συνοχή της κοινωνίας, όπως σας είπα προηγουμένως. Κάθε μεμονωμένος πολίτης, πιστεύω, έχει το δικαίωμα να προστατεύεται. Είναι κρίσιμο αυτό, να μπορούμε να προστατεύουμε τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο επίπεδο. Και γνωρίζω ότι υπάρχουν τομείς όπου θεωρούν οι πολίτες ότι στη γειτονιά τους δεν είναι τόσο ασφαλής όσο σε άλλες γειτονιές είτε λόγω προέλευσης, θρησκείας, χρώματος, φυλής. Δεν προστατεύομαι όπως κάποιοι άλλοι. Καμιά φορά έχει δίκιο και άλλοτε πάλι όχι. Όποιος σκέφτεται έτσι. Το οργανωμένο και το βαρύ έγκλημα. Πώς να το πω. Δεν πλήττουν μόνο τα συγκεκριμένα θύματα, αλλά και την ίδια τη συνοχή του κοινωνικού ιστού και αυτό είναι κρίσιμο. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τρόπο πολύ πιο αποτελεσματικό από ό,τι μέχρι τώρα. Γιατί αυτό δηλητηριάζει την κοινωνία. Αν οι πολίτες χάσουν την εμπιστοσύνη τους και πιστεύουν ότι δεν προστατεύονται ή με τον ίδιο τρόπο με άλλους πολίτες, τότε χάνεται ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της εμπιστοσύνης στην ίδια την κοινωνία, που είναι μεγάλο τμήμα της συνοχής. Αυτό το καιρό επεξεργάζομαι μια νέα στρατηγική ασφαλείας για την επόμενη πενταετία και φυσικά με μεγάλη χαρά θα ακούσω και τις προτάσεις σας γιατί τώρα ε, το, τις επόμενες εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα θα έχουμε τις νέες προτάσεις για τη στρατηγική αυτή. Το, ε, είπα, για το οργανωμένο και το βαρύ έγκλημα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη αντιμετώπιση και πιο αποτελεσματική από ό,τι στο παρελθόν θα πρέπει να τους εμποδίζουμε στο να βρίσκουν πυροβόλα, όπλα, εκρηκτικά και χρήματα. Τα χρήματα συνδέονται άμεσα με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύουμε τα εξωτερικά μας σύνορα καλύτερα, για λόγους ασφαλείας. Αλλά επίσης χρειαζόμαστε μια πολύ καλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία σε αυτό το τομέα. Έχουν εγκριθεί πολλά για τη διαλειτουργικότητα και θα πρέπει να εφαρμόζονται, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε. Ιδιαίτερα ότι ε, να πρόκειται για την προστασία των παιδιών, για την παιδική πορνογραφία, ε, την επιγραμμική. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κακοποίηση και η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Ε, η Ευρωπόλ κάνει πολύ καλή δουλειά και εντυπωσιακή σε αυτό το τομέα, αλλά θα πρέπει εμείς να κάνουμε πολύ περισσότερα. Είναι ευθύνη δική μας να προστατεύουμε τα παιδιά. επίσης να προστατεύουμε τα παιδιά από το τράφικινγκ, από τη διακίνηση, κορίτσια και γυναίκες. Χωράει βελτίωση μεγάλη εκεί. Επίσης είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ στη Χάγη τη Europol πριν αναλάβω καθήκοντα, αμέσως πριν, και εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Ε, όταν ήμουν εκεί είχαν μια πολύ μεγάλη κοινή δράση με ε, ηλεκτρονικές ψηφιακές πλατφόρμες και αστυνομικές δυνάμεις των κρατών μελών και με το FBI και ήταν μια πολύ επιτυχής κοινή δράση όπου ε, αφαίρεσε ε, τρομοκρατικό περιεχόμενο και έκλεισε σε μία νύχτα 26.000 λογαριασμούς στο διαδίκτυο. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Εκεί μπορούμε να προχωρήσουμε με θέληση, με θελοντική βέβαια συμμετοχή των ε, ψηφιακών πλατφορμών, αλλά χρειαζόμαστε και νέα νομοθεσία για να αφαιρείτε το τρομοκρατικό περιεχόμενο ε, στο διαδικτύο. Και ξέρω ότι αυτό το θέμα σας απασχολεί και σας. Επίσης θέλω να μιλήσω για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία ή evidence. Γνωρίζουμε τώρα ότι το 85% όλων των ε, έρευνών των αστυνομικών περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό είναι κρίσιμο και εδώ έχει σημασία πολύ κρίσιμη ο χρόνος. Πόσο γρήγορα μπορούν οι αστυνομικές διοκτικές αρχές που διεξάγουν τις έρευνες ε, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία που χρειάζονται για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο και το βαρύ έγκλημα. Πάντα φυσικά υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα ε, με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το σωστό τρόπο χρήσης ε, των νέων ευκαιριών. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να βρούμε ε, κοινέ λύσεις και να καταλήγουμε σε κοινά συμπεράσματα. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, με χαρά να τα συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε νέους δρόμους, νέους τρόπους για να προχωρούμε ε, και στο μέλλον. Να πω δύο λόγια και για τη μετανάστευση. Ασφάλεια και μετανάστευση είναι δύο στοιχεία του χαρτοφυλακίου μου. Και όταν τα συγκρίνω, υπάρχουν διαφορές στην εμπιστοσύνη. Στην εσωτερική ασφάλεια υπάρχει μεγαλύτερη ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη συνεργασία. Στη μετανάστευση, πιστεύω, χωλένουμε. Δεν υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών κατά την άποψή μου είναι ένας από τους λόγους αυτός που είναι τόσο δύσκολο να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Ναι. Καμιά φορά όταν υπάρχει αυτή η δυσπιστία ε, έχουμε πάρα πολύ λεπτομερή νομοθεσία και κανονισμούς. Καλύτερα να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία για το μεταναστευτικό. Αυτό θα είναι καλό. Και για αυτό το τμήμα του χαρτοφυλακίου μου να μην γίνονται οι συζητήσεις έτσι σε πολύ ψηλό επίπεδο και πολύ μεγαλόστομες δηλώσεις. Ε, να προσγειωθούμε λίγο. Ε, ε, γίνονται πολεμικές ανακοινώσεις περίπου, με πολεμικό λεξιλόγιο. Η μετανάστευση είναι κάτι που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Ο ρόλος μας είναι να διαχειριστούμε σωστά τη μετανάστευση και να την ελέγχουμε. Αυτό χρειαζόμαστε. Εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και φυσικά με το Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Στις ακροάσεις είπα ότι σκόπευα να κάνω διμερείς ε, συναντήσεις με όλα τα κράτη-μέλη πριν τα Χριστούγεννα. Τώρα όλο αυτό έχει ε, μετατεθεί κατά ένα μήνα μέχρι ε, τα τέλη Ιανουαρίου. Σε κάποιες επισκέψεις θα με ακολουθήσει ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και σε κάποια άλλα ε, θα είμαι μόνη μου με τα κράτη-μέλη. Τώρα κυκλοφορούν διάφορα non-paper. Ε, κάτι κινείται και δείχνει ότι τα κράτη-μέλη προσπαθούν να καταλήξουν σε μια νέα θέση. Και νομίζω καλό θα ήταν να αρχίσουν τα κράτη-μέλη να έχουν, πώς να το πω, μια εικόνα για το τι σημαίνει να είσαι στη θέση ενός άλλου κράτους μέλους. Διαφέρουν πάρα πολύ οι πραγματικότητες. Πέντε κράτη-μέλη επομίζονται το 90% ε, της παράτυπης μετανάστευσης ε, και 72% των αιτήσεων πηγαίνουν σε πέντε κράτη-μέλη τα οποία δεν είναι τα ίδια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 40 εκατομμύρια περίπου γεννιόνται σε τρίτη χώρα. Κάθε Δύο, 2-2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έρχονται να εγκατασταθούν ή να, ζήσουν για λίγο χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος θα έχουμε περίπου 100.000 παράτυπες διαλέψεις. Άντε, 120 ας πούμε, χιλιάδες. Ταυτόχρονα όμως θα έχουμε μάλλον 700.000 αιτήσει. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δευτερογενείς μετακινήσεις και είναι μεγάλο ζήτημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ε, προσπαθήσουν να πλησιάσουν τις θέσεις τους για να αλληλοβοηθούμε να βοηθηθούμε και πρέπει να σας πω ότι δεν θα ακούσω μόνο τα κράτη-μέλη αλλά και το Κοινοβούλιο και ξέρω ότι στην Επιτροπή σας σε κάποιες περιπτώσεις έχετε κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και πάρα πολύ εντυπωσιακή για τα θέματα αυτά. Ούτε θα αρχίσουμε από το μηδέν. Θα χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε όλη αυτή την προεργασία που έχει γίνει. Αλλά φυσικά θα πρέπει να γίνει και μια νέα κίνηση. Πότε θα είναι έτοιμο το νέο σύμφωνο, δεν ξέρω. Ε, Αλλιώ δεν θα είχε νόημα αν σα έδινα ημερομηνία να συζητήσω με τα κράτη-μέλη. Το σημαντικό, ένα από τα σημαντικό στοιχείο θα είναι η καταπολέμηση των διακινητών. Το δεύτερο, συνεργασία με τα, κράτη, τα τρίτα κράτη. Θα πρέπει να, βρούμε, να συνάψουμε εταιρικέ σχέσει και συνεργασίε με τα τρίτα κράτη. Και για να αποφύγουμε παράτυπε διελεύσει ανθρώπων που δεν είναι επιλέξιμοι για προστασία με το άσυλο, αλλά και να δημιουργήσουμε νόμιμους διάβλους να έρχονται οι άνθρωποι ε, και νόμιμα και έφτακτα να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στην οικονομία μας. Γιατί ο πληθυσμός μας γυράσκει, θα χρειαστούμε μετανάστες. Ε, πολύ σημαντικό λοιπόν είναι να συνεργαζόμαστε με τις τρίτες χώρες στην καταπολέμηση των διακινητών για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να βελτιώσουμε τη φύλαξη των συνόρων μας και να επιταχύνουμε τις επιστροφές. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στους πολίτες ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής σημαίνει ότι προστατεύουμε εκείνους που έχουν ανάγκη προστασία και υποδεχόμαστε επίσης εκείνους που θέλουν να εργαστούν και να συνεισφέρουν στην οικονομία μας. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να είναι ελεγχόμενα. Ποιος έρχεται και πότε. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές οι επιστροφές. Επίσης χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό αλληλεγγύης ε, και λόγω των γεωγραφικών ε, δεδομένων. πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Πώς ε, ε, χειριζόμαστε τις ε, μεταγκαταστάσεις, ή επανεγκαταστάσεις. Επίσης, κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Πρέπει να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό και τις διακρίσεις. Όσοι είναι επιλέξιμοι να ζήσουν στην Ευρώπη, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες, ε, είτε δικαιούνται. Είναι ευπρόσδεκτοι. Χαιρόμαστε που έρχονται εδώ και θέλουμε να επιτύχουν στη δουλειά τους, να κάνουν παιδιά, τα παιδιά τους να, να, μορφωθούν καλά και να έχουν ένα καλό μέλλον. Κοινωνία χωρίς αποκλεισμού. Καμιά φορά υπάρχει έτσι μια δευτερογενή τιμωρία στην οποία υποβάλλονται οι νέο αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο του νέου συμφώνου. Ήδη είμαι στα 10 λεπτά. Μόνο 10 λεπτά κάλυψα, τελείωσα. Thank you for making it 10 minutes because we... Ευχαριστώ που δεν ξεπεράσει τα 10 λεπτά γιατί έχουμε ένα μακρύ κατάλογο. Καταρχάς όσοι ήθιστε ή συντονιστές από κάθε πολιτική ομάδα. Δύο λεπτά έκαστος Και οι υπόλοιποι, μακρός οικοτάλογο, ένα λεπτό. Μια μισή ώρα έχουμε μόνο και έχουμε και την ψηφοφορία εν συνεχεία. Να εστιάσουμε λοιπόν στα όσα είπε η κυρία Γιωχάννησον και στα εκκρεμιστήματα. Κυρία Μετσόλα, έχει πρώτα το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Επίτροπη. Σας ευχαριστώ. Πολύ ξεκάθαρα λόγια. Και με ανυπαμονησία προσβλέπουμε στη συνεργασία μεταξύ μας τα επόμενα χρόνια. Θα εστιάσω στο πρώτο τμήμα της ομιλίας σας για την ασφάλεια. Η μέρα των Ηνωμένων κατά της διαφθοράς και φυσικά και δεν μπορώ να παραλείψω να αναφέρω τι συνέβη στη χώρα μου, τη Μάλτα. Η διαφθορά σκοτώνει. Έχει θύματα. 784 μέρες πριν ε, η δημοσιογράφος Ντάφνη Καρόνα Γκαλίτσια εκτελέστηκε έξω από το σπίτι της. Ένα από τα θέματα που έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια ήταν πώς μπορεί μέσω του συστήματος ε, ε, χορήγησης διαβατηρίου ε, έναντι μετρητών να αποτελέσει διάβλο προς την τρομοκρατία ή τα εγκληματικά κυκλώματα. Επί τόπου η κατάσταση παραμένει πολύ τεταμένη στη Μάλτα. Καθημερινά σχεδόν έχουμε διαδηλώσεις και σήμερα το πρωί μάλιστα που κατέλαβαν το γραφείο του Πρωθυπουργού Μουσκάτ, καλώντας τον διαδηλωτέ να παρετηθεί, γιατί ακόμα δείχνει αγκιστρωμένο ε, στην ε, έξωση. Αυτό που έγινε στη Μάλτα θα πρέπει να δράσει ως καταλήτης για να αναλυφθεί δράση ώστε αυτό το οποίο γίνεται σε ένα κράτος μέλος σήμερα να μην γίνει ε, ξανά στο μέλλον πουθενά. Τι γίνεται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε συναντηθεί, έχετε συνομιλήσει με τον αντίστοιχο Μαλτέζο ομόλογο ή τους ε, Μαλτέζους ομολόγους και τι προβλέπετε να κάνετε. Έχετε σχέδια να επικοινωνήσετε. Ευχαριστώ. Κυρία Σίπελ για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα μιλήσω για τη Μάλτα όχι γιατί διαφωνώ απόλυτα, ε, με κάποια τουλάχιστον πρόσφατα, αλλά γιατί παίρνει πολύ έντονο πολιτικό χαρακτήρα το όλο θέμα. Λοιπόν, που το λέω αυτό. Θέλω... It's true, <laughs> because there are many things we can talk about. Ναι, είναι αλήθεια αυτό γιατί πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος, παρακαλώ. Δεν έχουμε χρόνο. για να ασχολούμεθα με φήμες ή για να ακούμε ε, κάποιες ε, κραυγές ή επιφωνήματα από το κοινό. Ναι, αλλά βάλτε το χρονόμετρο στο μηδέν, πρόεδρε, γιατί μου φάγε χρόνο όλη αυτή η ιστορία. Ωραία. Δύο λεπτά λοιπόν έχετε. Επανέρχομαι, κυρία Ζήπελ, στα αποδεικτικά στοιχεία. Συμφωνώ απόλυτα με την Επίτροπο που είπε πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου Πρέπει ταχύτερα να ερευνούμε τα πράγματα. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που έγκυται στο γεγονός ότι τα δικαστικά και αστυνομικά συστήματα των κρατών μελών διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι όλοι οι σκιώδεις προσπαθούν να βοηθήσουν στην εξέβρεση λύσης για αυτό το πρόβλημα. Μιλήσατε για την ασφάλεια και την στρατηγική. Αναφερθήκατε επίσης στο γεγονό ότι σε μεμονωμένες ε, χώρες και ε, πόλεις υπάρχουν πολίτες που νιώθουν ε, περισσοτερο προστατευμένοι από άλλους σε άλλες πόλεις ή χώρες. Και αυτό αποτελεί πρώτα απ' όλα εθνική αρμοδιότητα τούτου λεχθέντος. Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει την εστίαση πρώτα απ' όλα στην εφαρμογή όλων όσων έχουν κατατεθεί ε, ως προτάσεις, γιατί πολλές φορές ε, σπέβδουμε να νομοθετήσουμε εκ νέου, όμως τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία πάντοτε και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τον καλύτερο έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων, συμφωνώ απόλυτα, διότι για παράδειγμα στη χώρα που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, Υπάρχουν όλο και περισσότερες ποσότητες ναρκωτικών και δικοκαίνης που μπαίνουν στη χώρα μας και θα έπρεπε να δούμε πώς γίνεται αυτό, πώς μπαίνουν στη χώρα μας και στις χώρες μας εν γέννη. Για τη μετανάστευση, το τελευταίο ερώτημα. Με ικανοποίηση άκουσα να λέτε ότι θέλετε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τις δευτερογενείς κινήσεις, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια. Σίγουρα πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα, να ανακόψουμε αυτά τα φαινομένα. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τουλάχιστον το υφιστάμενο πακέτο για το άσυλο. Αλλιώ δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο, και Ρέιν για την ομάδα Ρηνιού. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Επίτροπε, στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή μα. Αρχικά κάποιες παρατηρήσεις για το μεταναστευτικό σύμφωνο που περιμένουμε όλοι. σε συνέχεια τον όσο είπε Σίπελ. Ξέρετε ότι συνομιλούμε και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά πρέπει να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Το Κοινοβούλιο συνομοθετεί, είναι στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο. Άρα δεν δίνουμε κάποια συμβουλές, ψηφίζουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να πετάξετε έτσι στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτό είναι το νομικό ζήτημα, αλλά το 2015 αυτό το πακέτο ε, καταρτίστηκε ως απόπειρα να λυθεί ε, το αδιέξοδο που υπήρχε στο Συμβούλιο. Αυτό όμως δεν λειτουργήσε. Το ίδιο λάθος θα κάνουμε ξανά. Ξεκινώντας από το μηδέν, το πρόβλημα έγινε στο Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν και δεν αναλαμβάνουν ευθύνη. Δεν είναι πρόβλημα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για την ασφάλεια. Καταρχάς, προτού διατυπώσετε νέες προτάσεις ως Κομισιόν, γιατί δεν κάνετε αυτό που έχει ζητήσει ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη από το 2011, δηλαδή ενδελεχή αναλυτική αξιολόγηση όλων των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί είναι κάτι που ποτέ δεν έγινε, ποτέ. Πριν λοιπόν προτείνετε κάτι νέο, θα έλεγα καλύτερα να δείτε τι ήδη υπάρχει και αν αυτό χρειάζεται αλλαγές ή προσθήκες. Δεύτερον, νομίζω ότι το κράτος, το κράτος δικαίου σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι, αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας η Κομισιόν σε έναν βαθμό, αλλά κυρίω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα τελευταία ε, χρόνια έχουν λάμψει δια τη απουσία του. Και δεν νομίζω, κυρία Ζήπη, συγγνώμη, ότι έχει πολιτικοποιηθεί το θέμα τη Μάλτα. Εγώ ανησυχώ τα μάλα για το τι συμβαίνει. Και ιδίω για το γεγονό ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για να μπει η Ουγγαρία ε, δυσκολευτήκαμε πολύ. Για τη Μάλτα παλεύουμε. Η Πολωνία συζητήθηκε όχι σε Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό για την ασφάλεια της Υπήρου μας. Και είναι κάτι που η Κομισιόν πρέπει να το αντιμετωπίσει. Ευχαριστώ. Από τους to... Ευχαριστώ την κυρία Γιώχανσον που ήρθε να μας μιλήσει για πρώτη φορά και ε, με χαρά να συνεργαστούμε. Ε, σημειώνω αυτή την παρατήρηση για την ε, καχυποψία στη συνεργασία και τη διαφορά ανάμεσα στην αστυνομική συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια για τη μετανάστευση. αλλά σε πολλά κράτη-μέλη πραγματικά ε, επιδεινώνεται η κατάσταση του κράτους δικαίου και είναι πολύ ανησυχητικό. Για το νέο σύμφωνο για το άσυλο, για μας το σημαντικότερο ως αλλαγή ε, αυτό που χρειάζομαστε είναι να αλλάξει ο κανονισμός του Δουβλίνου. Έχουμε πολλή νομοθεσία για το άσυλο, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όντως με το Δουβλίνο και πραγματικά σας ε, παραπέμπω στην κοινή θέση του Κοινοβουλίου. Ε, νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Φυσικά περιμένουμε τις νέες προτάσεις σας. Ελπίζουμε να είναι αποτελεσματικές στην πράξη και να συνάδουν με την αρχή της αλληλεγγύης αλλά και τις αρχές ε, του κράτους δικαίου ε, και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο μεταξύ φυσικά ε, έχουμε πολλές ελλείψεις σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με το κεκτημένο του ασύλου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κοιτάξτε τι γίνεται στα ελληνικά νησιά, στα κροατικά σύνορα και πάει λέγοντας. Και ε, επανειλημμένα έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κοιτάξει και αυτό, να ε, συμμορφώνονται και να εφαρμόζουν την νομοθεσία τα κράτη-μέλη. Τι κάνετε εκεί κυρία Γιώχανσον και τι θα κάνετε και βραχυπρόθεσμα, εκθέσεις αξιολόγησης, ε, θα βγάλετε κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη για να συμμορφώνονται καλύτερα με τη χρηματοδότηση, τι γίνεται. Πιλωτικά προγράμματα, ξέρω εγώ, προσφυγές επί παραβάση, γιατί Υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων. Επίσης έχω πρόβλημα με την εξωτερική συνεργασία, με τον Ήγηρα, με τη Λιβύη, πολλά θέματα. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρες. Ε, η Επίτροπος υποσχέθηκε να το κοιτάξει και να δει και συστήματα ελέγχου για τη συμμόρφωση στις συμφωνίες αυτές. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι προτάσεις σας για αυτά. Από την ομάδα ID, Καρντίνο, όχι, αποσιάζει ε, εσείς, ο κύριος Σόφολτ. Κομισέ Ιουχένσον. Κύριε Επίτροπε, Είπατε για την μετανάστευση στην ακρόαση εκείνη που έγινε πριν οριστείτε επίτροπο, δεν εκπροσωπείτε την Σουηδία. Και υπήρχε μια εκπομπή ε, στην οποία βγήκατε πριν, ε, πριν την ακρόαση και είπατε ότι θέλετε να υπάρχει αλληλεγγύη υποχρεωτική και έτσι υποχρεωτικά να μοιράζονται οι μετανάστες. Ναι, και είπατε ότι είσαστε περήφανοι για την σουηδική μεταναστευτική πολιτική. Όμω και αλλού, στη Δανία α πούμε, κάποιοι δεν θέλουν ε, μετανάστε και εμεί θα δώσουμε αγώνα κατά αυτού. Ε, κατά αυτή τη πρόταση δηλαδή. Επομένω, δεν είναι λύση η σουηδική πολιτική, δεν είναι υποσχέσει ευρωπαϊκέ αυτέ. Είναι ένα πρόβλημα. Ο κόσμο προβληματίζεται πολύ για τη μετανάστευση και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει μια επίτροπο από τη χώρα που έχει την πιο ανεύθυνη μεταναστευτική πολιτική από όλες τις χώρες. Οπότε, εσείς, αφού θέλετε να συμβάλλετε στην πολιτική μετανάστευση, τελικά θα βοηθήσετε στο να έχουμε αυτό το τσουνάπι βιασμών και εγκλήματος από τις συμμορίες. Και έχω να σας προτείνω τα εξής τρία Κλείστε τα εξωτερικά σύνορα. Έλεγχοι στα ιστορικά σύνορα και να στείλουμε πίσω τους εγκληματίες μετανάστες. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος Προκατσίνη για το ECR. Να σας τα πω στα Ιταλικά. Συμπαθάτε με κυρία Γιώχανσον και σας ευχαριστούμε με αυτή την πρώτη ευκαιρία με την συνάντηση να σας ευχηθώ καλή δουλειά κυρία Επίτροπε. Δύο σημεία θέλω να θίξω, ασφάλεια και μετανάστευση. Για την ασφάλεια ήδη μας είπατε ότι είναι πιο δύσκολο να δούμε τι διαχωρισμοί θα γίνουν στο εσωτερικό. Κι όμως υπάρχουν, υπάρχουν διαφορές και διχασμοί όσον αφορά τη μετανάστευση. Και ας ξεκινήσουμε με τη σχέση ασφάλειας και μετανάστευσης, γιατί συχνά αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει αναφίβολα μια τέτοια συνάφεια και αυτό δεν οδηγεί σε κάποιο είδους ανάσχεση της λαθρομετανάστευσης, οπότε τελικά παραβλάπτεται και η νόμιμη μετανάστευση, κυρίως αυτή. Οπότε το μήνυμα που περνάει είναι ότι κανείς στην Ευρώπη μπαίνει μόνο παράνομα, πληρώνοντας ε, τους ε, διακινητές, ενώ μπορεί κανείς να μπει νόμιμα. Γιατί υπάρχουν οι ποσοστώσεις, αλλά τις έχουν εξαντλήσει τις ποσοστώσεις οι παράνομοι. Και σας ερωτώ. Πήγατε στην Τουρκία, ήταν η πρώτη σας ενέργεια μαζί με τον Επίτροπο Σχοινά, να δείτε τον Ερντογάν και τι θα λέγατε. Ποιο είναι το μήνυμα, τι βγαίνει από αυτή την συνάντηση, γιατί αυτό που με ανησυχεί είναι ότι συνεχίζει να πιστεύει ο κόσμος ότι η λύση είναι το να πασάρει στην Τουρκία τον έλεγχο. Τον έλεγχο των συνόρων γιατί δεν έχουμε το θάρρος να το κάνουμε αυτό οι ίδιοι. Ο πρώτος σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα για την ε, Γκουε. Κυρία Πελετιέ, εσείς είστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και κυρία Επίτροπε. Δύο λόγια για το σύμφωνο για τη μετανάστευση. Ανησυχούμε γιατί ο σκοπός είναι να περισταλούν τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο. Ε, δεν είναι εδώ να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο. Ε, επίσης, έχουμε την εντύπωση ότι αυτό το σύμφωνο που προτείνεται έχει σκοπό να εμποδίσει τη διακίνηση ε, και να παραβλάψει τα δικαιώματα. Εμείς θέλουμε κάτι να κάνετε, να αντιδράσετε όταν καταποτάνετε τα δικαιώματα των μεταναστών, των προσφύγων, των ετούντων, όταν αυτό δεν το κάνουν τα κράτη-μέλη και τους στέλνουν πίσω. Τώρα όσον αφορά αυτές οι επαναπροωθήσεις, τι γίνεται, για να πούμε για την Τουρκία. Αν ακούσουμε την Τουρκία σήμερα, έχουμε 340.000 οι οποίοι ε, γυρίζουν ε, εθελουσίως στην ε, Σύρια και έχουμε τις ΜΚΟ όπως τη Διεθνή Αμνηστία, το Human Rights Watch και ε, αυτές οι ΜΚΟ έχουν κάποια στοιχεία και λένε ότι δεν είναι και τόσο εθελούσια όλη αυτή η επιστροφή. Εφαίνεται ότι οι Τούρκοι τους ξεγελάνε, τους εξαναγκάζουν, ασκούν και δύο ακόμα τους βάζουν να υπογράψουν χαρτιά και να λένε εκεί να δηλώνουν θα γυρίσουν και ουσιαστικά αυτό γίνεται επομένω μια άσκηση βία. Αφού λοιπόν υπάρχει παραβίαση της αρχής μη επαναπρόθεσης, για πέστε μου. Δεν θα το πείτε αυτό στην Τουρκία ότι ανησυχούμε για αυτή την εξαναγκαστική επιστροφή που την μασκαρεύουν ως εθελούσια δεν θα πρέπει να σεβαστεί η Τουρκία την αρχή της μη επαναπροώθησης. Ευχαριστώ και συγγνώμη που έχω βραχνιάσει. Ευχαριστούμε και Πελέτη, αν την καλοσύνη κύριε Επίτροπε. Έχουμε πρόγραμμα να κάνουμε μια ψηφοφορία ή ηλεκτρονικά που δεν αργεί και πάρα πολύ. Οπότε θα πρέπει ευθύ αμέσω να πάμε στου υπόλοιπου συναδέλφου που έχουν κάτι να ρωτήσουν, γιατί έχω ένα τεράστιο κατάλογο από 25 συναδέλφου να ρωτήσουν. Ένα λεπτό, ένα λεπτό και όχι παραπάνω. Βοηθήστε, βοηθήστε και το καλό όλων. Και έτσι να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην ώρα μας. Ο κύριος Μωράης είναι πρώτος που θα λάβει το λόγο. Επίτροπε. Καλή επιτυχία όσον αφορά κυρίως το σύμφωνο. Και να σου πω την αλήθεια ότι υπάρχει πλούσια εμπειρία για τη Σουηδία και όταν λέμε για αλληλεγγύη, Μερικέ χώρε έχουν πιο αλληλεγγύη από άλλε. Αυτό ε, είναι θέμα τη Σουηδία. Ακόμα δεν έχετε κάνει τίποτα. Τι να σα ε, ε, ρωτήσω συγκεκριμένα. Όχι, όχι με την καλή έννοια το δεν κάνετε ακόμα τίποτα. Οπότε, δύο πραγματάκια σύντομα. Είπατε για αυτά τα non-paper, άρα έχουν ε, ενεργοποιηθεί τα κράτη-μέλη. Τι θα γίνει με αυτά τα non-paper, θα δοθεί το βάρος στις επιστροφές. Ε, βέβαια, θα πρέπει συνολικά αυτό να μπει στην πολιτική, αλλά τι είναι, κάποιο είδους προϋπόθεση, κάτι σαν αιρεσιμότητα, αλληλεγγύη, ε, νόμιμη είσοδος, ε, μπλε κάρτες. Για πέστε μας, τι θα κάνετε. Εσείς κύριε Ράντεφ έχετε τώρα το λόγο. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, Συγχαρητήρια και καλώς ορίσατε. Έχουμε αυτόν τον διαδρομένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας ενημερώνει η Επιτροπή και το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά ούτως ώστε να κάνουμε κάτι με τα προβλήματα της μετανάστευσης. Χρειάζεται επομένως κάτι επιγόντως να κάνουμε περισσότερα ή να κάνουμε κάτι για την Μεσόγειο γιατί τελευταίους μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες τραγωδιών στα ελληνικά νησιά. Η δε δήλωση ΕΕ Τουρκίας αποδίδει ακόμα, αλλά αυξάνεται η πίεση στην Τουρκία και υπάρχει φόβος αποστεροποίησης στην περιοχή. Με όλα αυτά τα δεδομένα, τι θα κάνει η Κομισιόν. Αυτή η αυξανόμενη πίεση δεν θα επηρεάσει το Σέγγεν. Όπως ξέρετε, Ακόμα υπάρχουν στερικοί έλεγχοι στα σύνορα Σέγγεν από κάποιε χώρε. Τι θα κάνετε, θα λάβετε τίποτε μέτρα, ο Πρόεδρος. Κυρία Σμάνη, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, συγχαρητήρια ε, για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Πολύ δύσκολο το έργο σας, όπως είπαν πολλοί προλαλήσαντες. Δύο ερωτήσεις. Είπατε προηγουμένως ότι θέλετε να έχουμε ασφαλείς και έφτακτες διαδικασίες για τη μετανάστευση. Είχαμε και ένα τεράστιο πρόβλημα με το τράφικινγκ, τη διακίνηση κοριτσιών και γυναικών που πέφτουν στα νύχια των οργανωμένων εγκληματιών. Το πρόβλημα είναι ότι η πρώτη τους επαφή με τη χώρα στην οποία ε, φτάνουν, μάλλον το πω αλλιώς, ο κανονισμός του Δουβλίνου τους υποχρεώνει να τις επιστρέφουμε στις χώρες ε, όπου μπήκαν για πρώτη φορά στην Ένωση, δηλαδή να πάνε στη χώρα του διακινητή. Ε, και μιλήσατε και για την υπόθεση αυτή του βιασμού στη Σουηδία. Οι περισσότεροι ε, ε, βιαστές ε, είναι Ευρωπαίοι εθνοτικά που βιάζουν γυναίκες και παιδιά. Όταν κατονομάζουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Πράγια. Ευχαριστώ πολύ. Μίλησατε για εμπιστοσύνη η εμπιστοσύνη των πολιτών, η, η άλλη εμπιστοσύνη ε, είναι κάτι σημαντικό για μένα και όχι να υποπτεύεται το ένα στον άλλο για εγκληματία. Και γι' αυτό μια από τι προτεραιότητε τη δική μου πολιτική ομάδας είναι η μαζική επιτήρηση να ε, τερματιστεί που σημαίνει ότι ε, παρακολουθούμε τους πάντες χωρίς να στοχεύουμε τις έρευνες σε ύποπτους για αδικήματα, για τέλη αδικημάτων. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι σύμφωνα με την ομολογία περί διατήρησης δεδομένων απόφαση του δικαστηρίου δεν θα προτείνει η Κομισιόν ένα ακόμη εργαλείο που θα προωθήσει ε, την ε, αδιάκριτη μαζική διατήρηση δεδομένων. Δεύτερη ερώτηση αφορά το θέμα της ασφάλειας. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ασφάλειας είναι το να νιώθει κανείς ασφαλής. Ανησυχώ λοιπόν γιατί πολλοί συμπολίτε μας δεν γνωρίζουν τους πραγματικούς κινδύνους από το έγκλημα. Σε κάποιους ε, τόπους μπορεί το έγκλημα να υποχωρεί, αλλά ο κόσμος που ζει εκεί από τα μίντια αποκομίζει την άποψη ότι ζει σε ένα πολύ επικίνδυνο μέρος και ότι ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι θα μπορούσατε ίσως να προτείνετε στο θεματολόγιο σας κάποια μέτρα που θα ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και θα τους κάνουν νιώθουν περισσότερο ασφαλείς. Κυρία Πιόρκ θα είχε τώρα το λόγο που δεν είναι όμως εδώ, άρα το λόγο θα πάρει ο κύριος... Α, ο κύριος Μπαρένα. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Συναντηθήκατε με τι ελληνικέ αρχέ την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλουμε να σα εκφράσουμε τι ανησυχίε μα. Πρώτα απ' όλα για το σχέδιο που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση ότι τα hot spot θα τα ε, ε, μετατρέψει σε κλειστά κέντρα, κλειστέ υποδομή χωρητικότητα 10-15 χιλιάδων. Ποια είναι η θέση τη Κομισιόν σε σχέση με αυτό το σχέδιο και θα χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για αυτά τα κέντρα κράτους ουσιαστικά στην Ελλάδα. Επίσης η πρόσβαση στο άσυλο ε, θα παρακολουθεί η νομική συνδρομή και συμπαράσταση, το δικαίωμα στην ε, έφεση, η ε, πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία. Υπάρχει το σχετικό νομοσχέδιο. Το συζητήσατε αυτό με την κυβέρνηση και επίσης ότι αφορά τη μετεγκατάσταση. Τι θα γίνει μέχρι να εγκριθεί το νέο Δουβλίνο παρακαλώ να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση από χώρες που χρειάζονται αλληλεγγύη, όπως είναι η Ελλάδα. Now it'll be... Κάνκο. εσείς. Εντάξει. Βέβαια, με βάση την ομάδα, την σειρά, εσείς θα έπρεπε να είστε πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώχανσον, λέει ο κύριος Φέστα. Μιλήσατε για την ε, ε, ανάγκη προστασίας, ε, την αίσθηση ασφάλειας και τα λοιπά. Όλοι έχουν το δικαίωμα του να νιώθουν ασφαλείς και θα πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα δεν δημιουργείται μόνο από την παράτη μετανάστευση αλλά και από την νόμη και είχαμε δολοφονία την προηγούμενη εβδομάδα ε, στην ε, ε, Γερμανία. Είχε λιβανέζικη υπηκότητα, αλλά ήταν νομίμως στη χώρα και αυτοί που έχασαν τη ζωή τους και στο εξωσφαρή ήταν αγγλικής υπηκότητας, αλλά με καταγωγή από μετανάστες. Αν λοιπόν η αίσθηση ασφάλεια είναι σημαντική για την κοινωνία, δεν θα πρέπει να πάψει αυτό το παγκόσμιο μεταναστευτικό ε, σύμφωνο να υποστηρίζεται και να ισχύει. Ευχαριστώ. κυρία Κάνκο. Κανκό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε κυρία Επιτροπέ και συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Θέλω να σας ρωτήσω για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Χρειάζεται οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την νομοθεσία που χρειάζεται για να υπάρχει και εμπιστοσύνη των πολιτών το επόμενο διάστημα, όχι μόνο την πενταετία και αργότερα, αλλά να προστατεύεται και ο κόσμος από το τράφικινγκ. Όπως είδατε τα τελευταία χρόνια δεν ακολουθούν τους κανόνες στα κράτη-μέλη, ούτε το μηχανισμό μετεγκατάστασης. Για να είναι όλα αυτά αποτελεσματικά θα πρέπει πάντες να τα εφαρμόζουν. Τι θα γίνει με αυτό το νέο σύμφωνο που σχεδιάζετε και για το οποίο μιλήσατε. Πώς θα καταφέρετε να εξασφαλίσετε ομοψυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούν όλοι τους κανόνες. Οποιαδήποτε νέα συμφωνία ε, πώς θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα διχάσει την Ευρώπη και θα φέρετε συγκεκριμένες λύσεις για αυτό το θέμα. Ο κύριος Πέτερς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα επανέλθω στο θέμα της ασφάλειας. Είπατε ότι η Ευρωπόλ έκανε καταπληκτική δουλειά και τονίσατε ότι στο μέλλον θα πρέπει να κάνετε περισσότερο να κάνουν για τα ναρκωτικά και για τις εγκληματικές οργανώσεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, το οποίο είναι το χρήμα. Ε, ο προπολογισμό της Ευρωπόλ και της Eurojust και άλλων οργανισμών. Πώς μπορείτε από τη μια να λέτε ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα και από την άλλη να μην έχουν τα απαραίτητα χρήματα στη διάθεσή τους. Δεν αυξάνεται η πρικοδότησή τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μορένο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Επιτροπό για την παρουσία της και πραγματικά συνεχίστε την περιοδία σας στις διάφορες πρωτεύουσες ακριβώς αυτή την προσπάθεια να αυξηθεί η εμπιστοσύνη για το μεταναστευτικό. Ε, ένα από τα κλειδιά είναι η αντίληψη που έχουμε για τη μετανάστευση. Δεν είναι πληγή, δεν είναι μάστιγα, δεν είναι απειλή, είναι πρόκληση, αλλά είναι και ευκαιρία, όπως είπατε και εσείς, είναι και αναγκαιότητα. Θα πρέπει ε, να μείνουμε σε αυτή την αίσθηση, ε, την αντίληψη. Στη συνέχεια, τα συνόδευτα ανήλικα είναι παιδιά, θύματα. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα στη Μεσόγειο ε, ε, ε, παραλίγο να γίνει τρομοκρατική απόπειρα σε ένα κέντρο υποδοχής στη Μαδρίτη. Παρακαλώ λάβετε το υπόψη. Έχουμε εδώ προτάσεις και εγώ προσωπικά. Μπορεί το θέμα να είναι εθνικό, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, διότι μας αφορά όλους και όλες. κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την πολιτική σας. Ε, ε, και στην ε, Σουηδία. Εγώ ήμουν δήμαρχος 30 χιλιόμετρα από το Καλέ και 15 χρόνια υποδεχόμουν εκατομμύρια πρόσφυγες και ποτέ δεν υπήρξε το παραμικρό φαινόμενο ε, παρανομίας και εγκληματικότητας. Τα hot spot ε, έχουν απάνθρωπες συνθήκες στα εξωτερικά σύνορα και κυκλοφορούν διάφορα non-papers που αναφέρατε που φαίνεται να θέλουν να ενισχύσουν την ευθύνη των κρατών μελών ε, για τα εξωτερικά σύνορα που κάνουν κλειστά κέντρα κράτησης και πολλαπλασιάζονται αυτά. Κινδυνεύει να εκτραπεί η κατάσταση. Τι σκέφτεστε γι' αυτό και θα μας βεβαιώσετε ότι το νέο σύμφωνο θα λαμβάνει υπόψη ε, τα δικαιώματα των μεταναστών και θα επιμερίζει ε, το φόρτο ακριβώς για να μην έχουμε δευτερογενείς μετακινήσεις. Ευχαριστώ κυρία Γιόντσαβα για ένα λεπτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο σας κύριε Επίτροπε. Πιστεύω θα κάνετε ό,τι μπορούτε, ούτως ώστε να πετύχετε. Πέρσι μιλήσαμε πάρα πολύ για το πρόβλημα της σημερινής πολιτικής ασύλου. Τα κρατημέλη πιέζονται και ε, χωρίς συμπαράσταση. Ρεαλιστικά θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στο μέλλον και σας ερωτώ. Ποιοι θα είναι οι βασικοί άξονες του συμφώνου το οποίο προτείνεται τι καινοτομίε θα θεσπίσετε τώρα για τη ε, διαφθορά. Ναι, η διαφθορά σκοτώνει, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε δύο δύο σταθμά, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η διαφθορά ε, υποσκάπτει την ε, δημοκρατία σε πάρα πολλές χώρες όπως και στην δική μου χώρα την Βουλγαρία που υποσκάπτει την ε, ελευθερία των ΜΜΕ και ούτε έρευνα δεν μπορεί να γίνει όσον αφορά την παρανομή μετανάστευση. Και πάλι σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας υποστηρίζουμε 100% αλλά μην ξεχνάτε ότι ο, ο χρόνος πιέζει και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ο επόμενος. Αγγελός Κόλλα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ε, όχι, δεν επιτρέπεται τόσος ενθουσιασμός. Συγκρατηθείτε. Κύριε Λόρνερ, ευχαριστούμε που ήρθατε και συγχαρητήρια για τα νέα καθηκοντά σας, δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα, χάρηκα που μου απαντήσατε στην ακρόαση ότι θα επικεντρωθείτε στα θέματα εμπιστοσύνη και συνεργασία των Μελών και όχι αναγκαστικά ε, θα έχετε καινούργια πράγματα, καινούργια ε, νομοθετήματα. Ε, και ξέρετε, ο κύριο Ντάμπερκ, ο υπουργό τη χώρα μου τη Σουηδία, είπε για, για νέο νόμιμα για κρατήσει. Και τι θα γίνει. Τώρα, στον αφορά το πολιτέ πλαίσιο, υπάρχει μια φιλανδική πρόταση. Έχουμε στην πολιτική ασφαλεία σημαντικέ περικοπέ. Θα υπάρξουν γιατί γύρω Europol, κατά τη γνώμη σα, αρκετά χρήματα. Πώ βλέπετε τι νέε προτάσει. Πώ θα εξασφαλίσετε η Europol και οι άλλε υπηρεσίε θα έχουν επαρκή χρηματοδότηση. Μάρκαρτ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και στην αρχή ήθελα να σα πω ότι είμαι και εγώ νέο μέλο στο Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχει μια πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο που τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται να καταφέρει να συζητήσει. Α πούμε, εγώ είμαι Γερμανό. Ότι τα περισσότερα εγκλήματα στη Γερμανία γίνονται από Γερμανού τεσσερα πέντε χρόνια δεν πρόκειται να το πει αυτό κανένας. Μόνο τα άλλα θα πει αυτή η ομάδα και ο νοήτο. Και ήθελα να ρωτήσω ακόμα, υπάρχει αυτό το non-paper από τη Γερμανία και σωστά είπατε ότι οι δευτερογενείς μετακινήσεις απασχολούν πολύ τους Γερμανούς, ιδιαίτερα τον Υπουργό Ιστορικών μας αυτή τη στιγμή. Και η απάντηση του non-paper είναι να τους αφαιρούμε τα δικαιώματα στα σύνορα, δηλαδή να μην υπάρχει νομική συνδρομή, να μην τους αφήνουμε να κάνουν τις αιτήσει για το άσυλο και να τους κλείνουμε σε κέντρα κράτησης. Εσείς είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό να λέμε στους ανθρώπους αυτούς ότι είναι ευπρόσδεκτοι και είναι στοιχείο της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Ε, πραγματικά είναι σωστό ε, άνθρωποι που ζητούν προστασία και εμείς να τους κλείνουμε σε κέντρα κράτησης. Ευχαριστώ κύριο Σντεχόφσκι. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα γενικά να μιλήσουμε εδώ όσον αφορά την ασφάλεια στις πόλεις και να φέρθηκε το καλέ. Σας ρωτώ, Επίτροπε, εσείς πώς το βλέπετε. συνεχίζουν και επιτίθενται στου φορτηγατζίδες. Καντάδες χιλιόμετρα μακριά από το καλέ γιατί θέλουν ε, οι διακινητές να στείλουν κόσμο αφού τον φορτώσουν κρυφά, του στείλουν στην Βρετανία. Τι θα γίνει. Το άλλη ερώτηση για τη Σουηδία. Με προβληματίζει η κατάσταση στη χώρα σας. Τι γίνεται με τα ρεπορτάζ του BBC News που δείχνουν ε, συμμορίες και άλλα πολλά. Εσείς κύριε. Βόλατ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στην ε, Επιτροπή κύριε Βόλατα, σα εύχομαι κάθε επιτυχία για το δύσκολο έργο σα. Βλέπουμε εικόνε στην Ευρώπη ε, αυτέ τι εβδομάδε και μήνε, πράγματα που δεν θεωρούσα εγώ ότι είναι δυνατόν να συμβαίνουν στην Ευρώπη, ιδίω σε ελληνικά νησιά και στα δυτικά Βαλκάνια. Ε, λόγω ακριβώ τη ε, κακή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση των τελευταίων ετών, για παράδειγμα, και στη Βοσνία έχουν γίνει σφάλματα. Εμεί όμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε όλα να τα εξωτερικεύματα πηγαίνουμε αλλού, ε, γιατί έχουμε ευθύνη και χρειάζεται μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και το δεύτερο, και άρρηκτα συνδεμένο με το πρώτο, για την ευρωπαϊκή στρατηγική δηλαδή, Πράγματι είναι προφανέ ότι χρειάζεται αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά από την άλλη πλευρά εξίσου σαφέ είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε και τα θεμελιώδη δικαιώματα στα εξωτερικά σύνορα. Και σίγουρα υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο, αλλά πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Ε, και δεν μπορεί οι σύνοριοφύλακες να αποφασίζουν ad hoc ε, αυτοί που είναι στα σύνορα, αν είναι παράτυποι μετανάστε ή ε, άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν διεθνού προστασία. Πρέπει να να βρούμε μία ε, σωστή νομική διαδικασία. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν εκ νέου παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Παρακαλώ όμως να σέβεστε όλοι το χρόνο. Είδα και εγώ που πήγα πρόσφατα στη Λέσβο την κατάσταση και πραγματικά είναι φρικτές οι συνθήκες ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα στοιχειώδη, τρόφιμα, φαγητό κτλ. Ε, είπατε ότι υπάρχουν κάποιες ε, εξελίξεις τελευταίες. Ε, φαίνεται ότι κλειστά κέντρα κράτηση είναι η λύση για την ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Στείλαμε στον Υπουργό Εστερικών επιστολή ζητώντα να αναλυφθεί δράση στην κατεπίκουσα αυτή ανθρωπιστική κατάσταση. Εσείς τι θα κάνετε για να βελτιώσετε τις συνθήκες διαβίωσης, να επιταχύνετε την επανένωση των οικογενειών για τα συνάδελφα παιδιά και ε, κατεπηγόντως ε, να γίνει μεταγκατάσταση για να λυθεί η κατάσταση επιτόπου γιατί πραγματικά εγώ ντρέπομαι που είμαι Ευρωπαίος ερετό, ερετός βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτη αυτή την εποχή. Μπαρτόλο ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στην προηγούμενη θητεία είχαμε βρει απάντηση στις σημερινές προκλήσεις και στη μετανάστευση. Αλλά τα κράτη-μέλη δεν κάνουν το ίδιο. Πέρασαν τρία χρόνια και πάνω, αλλά δεν μπορούσαν να τα βρούνε για το άσυλο. Και γνωρίζουμε ότι έχουμε αυτές τις προτάσεις που διτιμούνται και πάλι όσον αφορά τον κανονισμό του Δουβλίνου. Δεν συμφωνώ με το ότι αποσύρθηκε αυτή η πρόταση για τις προθεσμίες. Καινούρια πρόταση θα είναι το ίδιο φιλόδοξο όσον αφορά την ε, χώρα εισόδου. Χρειάζονται κάποια άλλα μέτρα που να καλύπτουν περισσότερους ε, και εκείνους που έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες. Τώρα όσον αφορά τη θάλασσα. Χρειάζεται ευρωπαϊκή προσέγγιση. Τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι η διάσωση ανθρωπιστική δεν θα ποινικοποιείται. Κύριε Θεοδωράκη, έχετε ένα λεπτό. Θα είμαι σύντομος. Επίτροπε. Συμβουλή και ερώτηση. Διοκτικές αρχές. Προβληματίζονται για το κατά πόσον ε, ε, στο θεματολογιό σας τις καλύπτεται. πυρογνώμονες, άλλα μέσα εφαρμογής του νόμου. Τι γίνεται με την ε, αξιόπινη χρήση της ε, πληροφορικής. Μίλησατε κι εσείς για πορνογραφία, και κλπ. Πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό το έγκλημα. Όταν πάντα στις πρωτεύους σας συμβουλεύω να πείτε στα κρατημέλη να σας βοηθήσουν, να σας δώσουν τα κρατημέλη τα μέσα να κάνετε κάτι όσον αφορά τις, ε, τις νόμιμες, τους νόμιμους διάβλους για τη μεταναστεύση. δεν γίνεται τίποτα. Μαγεία. Ο κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να αναθεωρηθεί, να κατευθυνθούν ιστορικοί σύνοροι. Τα είπαμε και το έκανα, είπαμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Να σταματήσουν οι παρανομίε στα ιστορικά και τα εξωτερικά σύνορα. Πήγαμε στην Ιταλία, στα σύνορα και από πρώτο χέρι είδαμε τι γίνεται με εκτοπισμένου και πρόσφυγε. Του αποθούν κάθε μέρα, Του στερούν τι βασικές ελευθερίες. Δεν λαμβάνουν υπόψη ότι είναι ευάλωτοι. Ασυνόδευτοι ανήλικοι. Αφήνονται στην τύχη του πού θα βρουν την προστασία. Μπορεί να επιληθούν ποινέ. Είδαμε όμω τι γίνεται από την Κροατία που είναι χώρα του Σέγγιν. Συγκεκριμένα, τι θα κάνετε. Πώ θα μπορέσετε να υπάρχει ένα έλεγχο ανεξάρτητο ούτω ώστε όλα τα κρατημέλη να συμμορφώνονται και να λειτουργεί η περιοχή Σέγγιν χωρί καταπάτηση δικαιωμάτων. Ένα λεπτό, κύριε Ρουίθ. Ευχαριστούμε που ήρθατε και ευχαριστούμε για όσα είπατε. Και συμφωνώ. 100%. Ιδίω με αυτό το οποίο είπατε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε ε, φιλοπόλεμη ρητορική όσον αφορά τη μετανάστευση. Σημαντικό. Αυτό που θα σα σας πω αφορά τι διαβουλεύσει με τα κράτη-μέλη. Ναι, είναι θετικό, όπως ελέγχεται, αλλά εάν πασίζεται για κάποια λύση ομοφωνία στο Συμβούλιο, αντί τη ε, πλειοψηφία κοντά στη θέση του Κοινοβουλίου, τότε κατεβάζουμε τον πύχη για τη συμφωνία που θέλετε για την μετανάστευση. Θα χαθούν πολλά στοιχεία όπως η κατάσταση. Κύριε Αντέλη. Ευχαριστώ. Λέει κύριο Αντέλη. Πολύ ωραία ότι κάνετε καινούργια αρχή. Γιατί όλοι αυτοί που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη κάνουν καμία τέτοια αρχή, τα βρίσκουν μπαστούνια. Γίνεται το ανάποδο και τι γίνεται με τα σύνορα της Κροατίας. Υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία. Το κράτος ασκεί βία. Ακλώνει τα στοιχεία. Τους επαναπροωθούν από εκείνα τα σύνορα οι Κροάτες. Τι θα κάνετε εσείς συγκεκριμένα. Πώς τους επαναφέρετε στην τάξη. Καταπατούν τα δικαιώματα. Να σταματήσει παρανομία. Ροβέρτη. Presidente, innanzitutto grazie signora Commissaria, <coughs> soprattutto ho apprezzato quello che lei ha detto a proposito dei... Πολύ ωραία μας τα είπατε για το τι χρειάζεται να έχουμε εταιρικέ συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Για την πορνογραφία και λοιπά. Είναι απίστευτο το φαινόμενο. Θα πρέπει οι ιδιωτικέ αρχές να εξειδικευτούν. Έχω να ρωτήσω τα εξή τρία. Πρώτον, συμφωνώ με τα θέματα που είπατε για την διαφθορά. Τι στρατηγία έχει η Κομισιόν, θα έχει στρατηγική κατά της διεθνούς διαφθοράς. Τι καινούργια μέσα πολιτικής θα ενεργοποιήσετε όσον αφορά τις συλλήψεις σε πραγματικό χρόνο στα σύνορα. Δεν γίνεται τίποτα τώρα. Ούτε η Κομισιόν, ούτε το Κοινοβούλιο λένε τίποτα. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε για το, το οργανωμένο έγκλημα με επιτάξεις και κατασχέσεις για κάποια πολιτιστικά αγαθά. Τρίτον, συμφωνείτε με αυτό που πρόσφατα κατέβασε η προηγούμενη Κομισιόν για διάφορες τράπεζες που δεν σέβονται την ανακύκλωση. Θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκό όργανο και να εξασφαλίζει το ότι αυτού του είδους η ανακύκλωση θα απαγορεύεται και θα διώκεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε. Συγχαρητήρια για τον ορισμό σας. Σας περιμένει δύσκολη δουλειά, περίπλοκη λέει η κυρία Φεράρα. Τώρα όσον αφορά την ασφαλεία είπατε ότι είδατε ότι υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη των κρατών μελών, όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την ανταλλαγή των στοιχείων και έτσι υπάρχει περισσότερη ασφάλεια στην κοινότητα. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε τις νομικές βάσεις, τις νομικές διατάξεις που θα μας ασφαλίσουν περισσότερη ασφάλεια και εδώ εννοώ την διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την νομοθετική πρωτοβουλία του 16 όσον αφορά το να γίνει ευρωπαϊκό έγκλημα η σύσταση συμμορίας μαφίας. Επίσης, είπατε για fresh start. Τις πιστώ γιατί θα πρέπει να σταματήσει η αδράνεια. Αλλά το κοινοβούλιο έκανε πάρα πολλά και ήμουν εγώ η συγγήτρια για τη σχετική έκθεση. Μεγάλες οι προσπάθειες που έγιναν για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο να εγκριθεί. Καθυστέρησε. Μια νέα πρόταση και αυτή μπλοκάρεται. Σήμερα είχαμε 55 μαθητές που έκαναν επίσκεψη και με ρωτήσανε τι κάνει η Ευρώπη, τι κάνει για τη μετανάστευση και αναγκάστηκα βέβαια να τους πω την πικρή αλήθεια. Κυρία Κινίτσε, ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, ευχαριστούμε που ήρθατε. Συμφωνώ με όσα είπατε για την εσωτερική ασφάλεια θα πρέπει να αναβαθμίσουμε συνεργασία και περισσότερη εμπιστοσύνη των κρατών μελών. Ναρκωτικά, δουλεμπόρια, τα πιο βαριά εγκλήματα θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και τη διαφθορά που είπατε. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν μαφίες πίσω από τέτοια εγκλήματα. Εσείς δεν συμφωνείτε ότι ήρθε η ώρα να χαράξουμε ενιαία στρατηγική στην Ευρώπη για να ανασχέσουμε τις μαφίες. Έγινε αυτό στην προηγούμενη θητή για την ε, τρομοκρατία. Να εξυγχρονίσουμε τον ορισμό της σύστασης ε, μαφιός και συμφορίας. Τώρα έχει ξεπεραστεί το σχετικό νομοθέτημα που υπάρχει για τους ανήλικους μετανάστες, τα είπαν οι συνάδελφοι, αλλά η πλειοσύνη των ανηλίκων είναι κάτι που με απασχολεί γιατί έχουμε ένα ψήφισμα για την 30η επέτειο της σχετικής σύμβασης του ΟΗΕ και είπαμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κέντρο για να καταπολεμήσουμε την εκμετάλλευση και άλλα εγκλήματα κατά των ανηλίκων όταν έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Τι λέτε γι' αυτά? Ελπίζω να μην ξεχάσετε και κανείς να ε, πήρατε όλοι το λόγο. Δεν ήταν απορία άξιο που ζήτησαν τόσο πολύ το λόγο. Κυρία Επίτροπε, να το περιμένετε αυτό, να το έχετε υπόψη σα. Ξέρω ότι δεν είναι καλύτερη μέρα, είναι Δευτέρα απόγευμα. Παρ' όλα αυτά, όποτε και να έρχεστε για συζητήσεις, θα γίνονται συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή μας. Σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, συμπαθάτε με λίγο χρονικά. Ε, είχε προγραμματιστεί η ψηφοφορία να αρχίσει ε, σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, να αφήσουμε 20 λεπτά στην κυρία Πίτροπο για να απαντήσει, γιατί 25 ερωτήσεις έγιναν, εκτός από τους συντονιστές. Να τη δώσουμε ένα 20 λεπτό και μετά θα ακολουθήσει σύντομη ψηφοφορία, ε, τελειώσουμε. Βέβαια μετά έχουμε και συνεδρίαση των συντονιστών. Και παρακαλώ όσοι θέλετε να παραμείνετε στη συνεδρίαση των συντονιστών, μην φύγετε. Οι υπόλοιποι ε, μπορεί να φύγουν. Είναι πολύ σύντομη η ψηφοφορία. Τρεις ε, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες θα κάνουμε. Οπότε ας έχει λίγο χρόνο περισσότερο η Επίτροπος για να κάνει ό,τι μπορεί και να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που έγιναν. 20 λεπτά για να ε, συνοψίσετε τις ε, σκέψεις σας και να μας τις παρουσιάσετε. Έχετε το λόγο κυρία Πίτροπε. Ευχαριστώ. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις πολύ καλές ερωτήσεις αλλά και τις σκέψεις των ε, βουλευτών για τη μελλοντική νομοθεσία και χάραξη πολιτικής και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ορισμένε ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, με ανησυχεί ιδιαίτερα ε, η Μάλτα και η πρόσφατη κατάσταση και οι τελευταίες εξέλιξεις εκεί. Πρέπει σίγουρα να καταδικαστεί απερίφραστα η δολοφονία και πρέπει να πω ότι η Europol είχε κομβικό ρόλο στο ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ έρευνα που σημαίνει ότι η Europol είναι προστέμενη αξία για την επίλυση πολύ, πολύπλοκων και σημαντικών υποθέσεων και τη διαλεύκανσή τους. Η διαφθορά έχει θύματα ανθρώπινες ζωές. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. σε ό,τι αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο συμβουλίου. Η αντιπρόεδρος Βέρα Γιούρεβα και ο Επιτρόπος Διτιά Ρέιντερς είναι αυτοί που είναι αρμόδιοι για το κράτος δικαίου και σίγουρα θα συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση. Για την κυρία Ζήπελ, πράγματι είναι ε, πολύ σημαντική εφαρμογή. Πολλές αποφάσεις έχουν ληφθεί που πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα το να παρακολουθώ κατά πόσον πράγματι εφαρμόζονται οι αποφάσεις. Αλλά θεωρώ ταυτόχρονα ότι είναι αναγκαίες και κάποιες προτάσεις για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Για την κυρία Ιντβέλτ, ε, φυσικά και δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν, το έλεγα πάντοτε αυτό, ότι μπορούμε αυτές τι προτάσεις που είναι επιτάπητο και το σημαντικό έργο που έχει ήδη γίνει πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Υπάρχουν όμως δύο συνομοθέτες και χρειάζονται και δύο. Η κατάσταση αυτή είναι δύσκολη. Κάθε εβδομάδα που δεν έχουμε κοινό σύστημα κοινή πολιτική, κοινού κανονισμούς για το άσυλο και τη μετανάστευση, το τίμημα είναι υψηλό. Πολύ υψηλό κατά την άποψή μου. Το πληρώνουμε σε ό,τι αφορά την έλλειψη συνοχή και εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, αλλά το τίμημα το πιο υψηλό το πληρώνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που είναι εγκλωβισμένοι και στιβαγμένοι ε, στις διάφορες δομές στα ελληνικά νησιά και αλλού. Είναι παραδειγματικά κατεπίδουσα κατάσταση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε χωρίς να ξεκινάμε ταυτόχρονα και από το μηδέν. Δεν είναι κάτι που θα άρεσε κανέναν. Πρέπει δηλαδή να ενισχύσουμε τα όσα ήδη γίνονται. Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική αλληλεγγύη, είναι αδύνατο, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, να κατατεθεί στη, στο επίπεδο συμβουλή μια πρόταση με την οποία θα συμφωνήσει η πλειοψηφία ή τόσο θα υπάρξει συνένεση, ομοφωνία. αν δεν υπάρχει υποχρεωτική, ή μάλλον αν υπάρχει το στοιχείο της υποχρεωτικής αλληλεγγύης της μεταγκατάστασης. Σίγουρα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των χωρών πρώτης ε, εισόδου. Για τις ε, συνθήκες στην Αθήνα, κυρία Στρίκ, ήμουν και εγώ μαζί με τον Αντιπρόεδρο ε, Μαργαρίτη Σχοινά Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό και με τους άλλους αρμόδιους υπουργούς και για μένα ήταν ε, μια ευκαιρία να συναντήσω και ΜΚΟ, από τις οποίες αποκόμισα πολύ σημαντικές πληροφορίες επίσης και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν πως κατάσταση σε καταλυσμούς όπως αυτό της Μόριας είναι απαράδεκτες και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια τομή θα παρακολουθούμε την εφαρμογή της νέας ε, ελληνικής νομοθεσίας ε, και όταν μίλησα με τις ΜΚΟ και τις ρώτησα ποια είναι η άποψή τους για αυτή τη νέα νομοθεσία. Αυτό που τόνισαν είναι ότι θα μπορούσε να είναι κάτι καλό ή κακό ανάλογα με την εφαρμογή, το πώς θα εφαρμοστεί. Αυτό ε, θεωρούν το πιο σημαντικό. Είναι κάτι που έμαθα από αυτές. Την Κεσόφολτ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για, ε, με τη φρασιολογία που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για τους ανθρώπους. Ε, μην χρησιμοποιούμε λέξεις ε, που παραπέμπουν ε, σε θαλάσσιες καταστροφές, τσουνάμι κτλ. Μιλάμε για ανθρώπινα όντα και όλοι έχουν την ίδια αξία. θα ήταν πιο εύκολο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ε, μάλλον θα ήταν εύκολο να προχωρήσουμε σε μια λύση αν προσέχουμε περισσότερο τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Πολλές, πολλές ερωτήσεις. Πολλοί ρώτησαν πώς θα είναι αυτό το νέο σύμφωνο. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι στην σαουκή μου παρέμβαση σας έδωσα κάποιες αδρές γραμμές ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία αυτού του συμφώνου. Σίγουρα πρέπει να ακούσουμε όμως εσάς και τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να καταθέσουμε μία πρόταση η οποία δεν θα ε, περάσει, δεν θα λειτουργήσει. Σε ό,τι αφορά τα διάφορα επίσημα έγγραφα, τα non-paper, ε, δεν ε, έχω να πω πολλά. Τα κράτη-μέλη με αυτά τα non-paper ουσιαστικά θέλουν να δουν αν πετάει ο γάιδαρος. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τα πόδια μας ε, στη γη. Θα τα μελετήσουμε κάποια από αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι θέμα ασφάλειας. Αλλά σχετίζεται και με τις ε, διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται στα σύνορα για όσους έτουνται άσυλο. την κυρία Αλσαχάν. Ναι, τώρα μιλάω ε, σου ειδικά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε κατά νου ότι πολλά από τα παιδιά που φθάνουν είναι θύματα. Κάποια είναι, ε, έχουν ε, πέσει θύμα διακινητών. Κάποιοι βέβαια μπορεί να λένε ότι ανήκουν σε κάποια οικογένεια και να μην ανήκουν και άλλοι μπορεί να λένε ότι είναι ανήλικοι ενώ δεν είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τους νέους, τα παιδιά να τους ε, πάρουν πολύ στα σοβαρά όταν φτάνουν στα σύνορα και να υπάρχει στα σύνορα μια διαδικασία ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Για να μην έχουμε τελικά θύματα για μια ακόμη φορά θύματα κλιματικών δικτύων, γιατί ήδη ήταν αντικείμενο διακίνησης πολλά από αυτά τα παιδιά και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ξαναπέσουν στα νύχια ε, τέτοιων διακινητών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Europol, στα αγγλικά πάλι, δεν ξέρουμε ε, αν θα έχει επαρκή χρηματοδότηση, γιατί είναι υποσυζήτητο το πια αυτή τη στιγμή. Όπως και εσείς, έτσι και εγώ, γνωρίζουμε ποιες είναι οι διάφορες προτάσεις σίγουρα επηρεάζεται ο προϋπολογισμός της ασφάλειας. Έχουμε δει τι προτάσει τη Συνάδελφη Προεδρία, για παράδειγμα. Πάντω, σίγουρα θέλουμε να υπάρχει παρκές χρηματοδότηση για ε, πολύ σημαντικά αυτά καθήκοντα τη Europol. Για να δω. Με ικανοποίηση άκουσα να λένε ότι δεν μιλάμε για εμπιστοσύνη μόνο μεταξύ κρατών μελών, ε, αλλά και μεταξύ των πολιτών. Πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική και συμφωνώ. Αλλά επί του πρακτέου ε, για τη διατήρηση δεδομένων. Εγώ νομίζω ότι νομοθεσία χρειάζεται για τη διατήρηση δεδομένων. Έχουμε κρεμίσει υποθέσει στο δικαστήριο και δεν μπορώ, είναι πολύ νωρί τώρα, ε, δεν μπορώ να καταλήξω σε συμπεράσματα. Πρωτού δω την έκβαση αυτών των υποθέσεων, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση αυτή τη στιγμή. Νομίζω αυτά είχα να πω. Θαυμάσια. Είχατε περισσότερο χρόνο, αλλά δεν τον εξαντλήσατε. Ήταν ένας πρώτος γύρος ερωταπαντήσεων. Καλή αρχή. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερα να διαφωνήσουμε και σίγουρα περιμένουμε να έχουμε και άλλες ευκαιρίες αργότερα για να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο. Γιατί αξίζει δεν ναι, τα συζητούμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε για αυτό τον πρώτο διαρθρωμένο διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως σας είπα, σας παρακαλώ να παραμείνετε στην αίθουσα για να ψηφίσετε. Είναι μικρή η ψηφοφορία. Τρία πατήματα κουμπιού είναι ηλεκτρονικά και τελειώσαμε. Stay in the room Και να μην φύγουν οι συντονιστές. Και φυσικά να έχετε τις κάρτες σας ε, ψηφοφορίας. Now, electronic cards. Get them ready. Παρακαλώ, ετοιμάστε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε. Θα είναι γρήγορη ψηφοφορία. It can be fast. Okay. Now. Let's proceed. Λοιπόν, προχωρούμε. Ψηφίζουμε. First of all, we are... Πρώτη ψηφοφορία. Σχέδιο σύστασης. Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας κριτήρια και μηχανισμοί καθορισμού του κράτου που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχή ασύλου που υποβάλλεται σε κράτο μέλο ή στην Ισλανδία ή την Ορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολή του νόμου. Η συγκήτρια κυρία Βυσνιεύσκα. Είναι σχέδιο σύσταση, Η κυρία Βυσνιεύσκα απουσιάζει γιατί είναι σε αποστολή στην COP25 στη Μαδρίτη. Ψηφίζουμε λοιπόν παρόλα αυτά το σχέδιο σύσταση. με ονομαστική κλίση για το σχέδιο ψηφίσματος. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με μεγάλη διαφορά, δύο ψήφοι κατά χωρίς αποχές. Δεύτερη ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα των διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοφυλακή και Εκτοφυλακή. Άρχεται η ψηφοφορία με νομαστική κλίση και αυτή. Η συγκεκριμένη είναι η κυρία Ρομπέρτα Μετσόλα. Σκιώδης η κυρία Μαρίνα Κάλιολαντ. Λοιπόν, πάμε. Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις οργανικές διαπραγματεύσεις. Πέρας. Με την ίδια πλειοψηφία. 46 υπέρ, 2 κατά. Εγκρίθηκε. Και τώρα, η τελευταία ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα τη προσωρινή συμφωνία που προέκυψε από τι γερμανικέ διαπραγματεύσει σχετικά με τον κανονισμό για τι κοινοτικέ στατιστικέ για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Η συγητής είναι ο Γιάνν Κριστόφ Ότιεν και ο Πιέτρο Μπαρτόλο Κιώδη. Ψηφίζουμε τώρα. And the vote is closed. Πέρας. Και πάλι 47 υπέρ. Κανείς κατά μία αποχή. Ευχαριστώ πολύ. Λήξεις. Παρακαλώ να παραμείνουν οι συντονιστές. Ευχαριστώ. Presidente.